και έχει διδάξει κατά το παρελθόν σε μία σειρά πανεπιστημίων. Έχουμε λοιπόν εμπειρογνώμονες που πραγματικά έχουν επενδύσει επαγγελματικά τη σταδιοδρομία τους ε, στην ευρύτερη κατανόηση ε, των δημοψηφισμάτων ως ε, δημοκρατικού εργαλείου. Προτείνω λοιπόν πρώτα να δώσουμε το λόγο στους συντάκτες της μελέτης ε, που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στους ε, δόκτωρες ε, Μάριο και Φερνάντο Μέντες. Παρακαλώ, όποιος θέλει να πάρει το λόγο, πρώτος. μελητή. Is that right? Yes, thank you. Ευχαριστώ. Θα ξαναξεκινήσω. Αγαπητή Πρόεδρε, αγαπητά αξιότιμα μέλη, ο κύριο ε, Μέντε και εγώ με τα χαρά βρισκόμαστε εδώ στην σημερινή συνεδρία για να σα παρουσιάσουμε την μελέτη μα για τα δημοψηφίσματα επί ευρωπαϊκών ζητημάτων. Η παρουσίασή μα ε, θα ακολουθήσει ουσιαστικά τη δομή τη ε, μελέτη αυτή καθ' Θα παρουσιάσω τα τμήματα 1 και 2, 7 και 8. Και ο δεύτερο συντάκτη θα παρουσιάσει τα τμήματα 3 και 6. Δύο λόγια αρχικά για την στάθμιση της άμεσης δημοκρατίας ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά έχουμε τρεις κατηγορίες ε, ε, άμεσων δημοκρατιών. Αρχικά έχουμε ένα δημοψήφισμα σε ευρωπαϊκό ζήτημα, το οποίο διεξάγεται είτε από κράτος μέλος, είτε από, ένα, από μια περιφέρεια, Ενό κράτου μέλου. Μετά έχουμε πρωτοβουλίε πολιτών που διεξάγονται σε επίπεδο κρατου μέλου για ένα ευρωπαϊκό ζήτημα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει και σε δημοψήφισμα σε ορισμένε περιπτώσει. Είχαμε βέβαια και το επίμαχο πρόσφατο παράδειγμα ε, του δημοψηφίσματος στις κάτω χώρε για την Συμφωνία Σύνδεσης με την Ουκρανία και μετά έχουμε και ε, το, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ε, που είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια πρωτοβουλία άμεσης δημοκρατίας. Από πλευρά σύγκριση δεν έχει νόημα να εξετάσουμε του διεθνεί οργανισμού, γιατί κανένα από αυτού του οργανισμού δεν ε, παρέχει λειτουργίε άμεση δημοκρατία. Και μόνο σε πολύ σπάνιε περιπτώσει αποτελούν το αντικείμενο τέτοια χρήση άμεση δημοκρατία. Για του σκοπού τη μελέτη, λοιπόν, εξετάσαμε ε, εν συντομία μία συγκριτική ομοσπονδιακή προσέγγιση. Εδώ, λοιπόν, βλέπουμε στην βιβλιογραφία ότι ε, μεταξύ των ε, δημοκρατικών ομοσπονδιών ε, τα δημοψηφίσματα σε ομοσπονδιακό επίπεδο προβλέπονται, όμως η χρήση τους, με την εξαίρεση της Ελβετίας πιο συγκεκριμένα, είναι αρκετά σπάνια. Αν δούμε τώρα την δυνατότητα άμεσης δημοκρατίας από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή με πρωτοβουλίες πολιτών για ομοσπονδιακά ζητήματα, και αυτό είναι αρκετά σπάνιο ακόμα και στις πρωτοβουλίες θεματολογίου που θεωρούνται πιο ε, ήπιες. Και αν εξετάσουμε τα ε, δημοψηφίσματα κατόπιν πρωτοβουλία πολιτών, είναι και πάλι σπάνιο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο το βρίσκουμε μόνο στην Ελβετία. Εξετάζοντα λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση από συγκριτική ε, άποψη, μπορούμε να πούμε ότι στην ουσία η πρωτοβουλία των πολιτών είναι ένα αντίστοιχο επίτευγμα γιατί παρέχει διόδους ε, της για άμεση συμμετοχή των πολιτών ε, για κάτι το οποίο είναι το αντίστοιχο ε, ενός ομοσπονδιακού ζητήματος. Τώρα, σε ό,τι φορά τις κατηγορίες που έχουμε προσδιορίσει, αρχικά έχουμε ε, ένα, μια τετραπλή δέσμη ευρωπαϊκών δημοψηφισμάτων. Αρχικά έχουμε τα δημοψηφίσματα για την ένταξη, προσχώρηση κυρίως και ουσιαστικά όλα τα κύματα της ευρωπαϊκής διεύρυνσης ε, εκτός ε, της νότιας διεύρυνσης που έγινε το 1980, όλα τα υπόλοιπα λοιπόν οδήγησαν σε δημοψηφίσματα ε, ένταξης από τα υποψήφια προς ένταξη κράτη-μέλη. Μετά έχουμε και μια άλλη κατηγορία για την αποχώρηση. Μόνο ένα κράτος μέλος, το Ηνωμένο Βασίλειο πρόσφατα διεξήγαγε τέτοιο δημοψήφισμα για την αποχώρηση ε, της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά ε, τα δημοψηφίσματα για την αναθεώρηση των ε, συνθήκων έχουν ε, χαρακτηρίσει κάθε μεγάλη περίοδο αναθεώρησης της συνθήκης. αν δούμε ποιε χώρε έχουν διεξαγάγει ε, τέτοια δημοψηφίσματα, βλέπουμε ουσιαστικά πρόκειται μόνο για έξι κρατημέλη και τα περισσότερα εξηγούνται από τις ε, συγκεκριμένες συνταγματικές ε, περιστάσεις Ιρλανδίας και Δανίας. Μετά έχουμε και τα δημοψηφίσματα πολιτικής, κυρίως το δημοψήφισμα διεύρυνσης που έγινε στη Γαλλία την δεκαετία του ε, γιατί στη Γαλλία προβλέπεται στο Σύνταγμά της ε, μια συνταγματική ε, κλίδα σε ό,τι αφορά την πιθανή μελλοντική διεύνηση. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει περαιτέρω διεύνηση. Και τέλος, έχουμε και τα δημοψηφίσματα των τρίτων χωρών που διεξάγονται κατά κύριο λόγο στην Ελβετία δηλαδή χώρες που δεν είναι υποψήφιες ε, για ένταξη. Αυτές είναι οι τέσσερις κατηγορίες. Μετά, δεύτερη κατηγορία, έχουμε την λογική για την διεξαγωγή τέτοιων ε, δημοψηφισμάτων. Αρχικά έχουμε δημοψηφίσματα για σκοπούς συνταγματικότητα. Εδώ έχουμε το προφανές παράδειγμα της Ιρλανδίας. Μετά για ε, λόγους ε, κυρίως ε, τα δημοψηφίσματα που αφορούν την ένταξη ε, διέπονται από αυτή τη λογική και μετά έχουμε και άλλα δημοψηφίσματα για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας όπως ε, είναι το δημοψήφισμα του François Μιτεγόν στις αρχές του 1990 για την συνθήκη του Μάστριχτ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον συναδελφό μου για το τμήμα 3. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, θα σας δείξω κάποια γραφήματα τώρα. Πρώτα απ' όλα την κατανομή ε, των ε, δημοψηφισμάτων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Έχουμε αποκλείσει από τη συγκεκριμένη έρευνα της, τα δημοψηφίσματα των τρίτων χωρών. Γι' αυτό λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι έχουμε 48 δημοψηφίσματα

Ε, εκ των οποίων τα μισά ε, περίπου αφορούν το θέμα της ένταξης, αλλά ε, επίσης και τις τροποποίησης των συνθήκων. Εάν δούμε την κατανομή κατά λογική, θα δούμε ότι υπάρχουν πολλά δημοψηφίσματα τα οποία αφορούσαν κομματικά ζητήματα ή ζητήματα από των οποίων κάποιος θα έπρεπε να πάρει θέση. Αν δε ε, και την περαιτέρω λογική, καταλαβαίνετε εδώ, ε, ο, τον κατακαιρματισμό. Ε, ο πρώτος, η πρώτη στήλη που αφορά ε, τα δημοψηφίσματα ε, για την ένταξη, αυτά έχουν γίνει για λόγους ιδιοκτησίας κυρίως, ενώ αυτά τα οποία αφορούν την συνθήκη είχαν τη λογική της συνταγματικότητας. Ε, ακόμα είναι πολύ νωρίς ε, για να δούμε πώς αυτού του είδους ε, τα δημοψηφίσματα μπορούν να έχουν επίπτωση στη γενικότερη κατάσταση. Βλέπουμε εδώ τα δημοψηφίσματα για ένταξη με κόκκινο και τα υπόλοιπα με πράσινο. 80% των δημοψηφισμάτων ε, ε, είχαν ε, μάλλον αρνητικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι ένα νέο φαινόμενο. Περίπου ένα τρίτο των δημοψηφισμάτων έχουν αρνητική εξέλιξη. Ε, απ' την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι περίπου ε, ένα τρίτο ε, αποτυγχάνουν ασχέτως του θέματος. Εδώ βλέπουμε ένα, μια, ένα γράφημα το οποίο δεν είναι πάρα πολύ καθαρό αλλά δείχνει ότι υπάρχει, υπάρχουν δεκαετίες η γραμμή του χρόνου στο κάτω μέρος του γραφίσματος του γραφήματος ε, και ε, ε, έχουμε λοιπόν και με μία πράσινη γραμμή το όριο του 50%. Βλέπετε λοιπόν ότι έχετε εδώ πολλές γραμμές, πολλές, πολλά σημεία κάτω από τη γραμμή του 50%. Πριν από το 2000 περίπου ένα τέταρτο των δημοψηφισμάτων απετύχαναν και αυτό το ποσοστό ανεβαίνει στο 48% 100, κυρίως μετά από το 2010, ε, δηλαδή όταν ξεκίνησε η μεγάλη κρίση, ε, βλέπουμε ότι το ποσοστό φτάνει στο 60 και ξεπερνάει το 60%. Ε, ας δούμε τώρα δύο αυτές τις δύο διαστάσεις οι οποίες εξηγούν ή αιτιολογούν αυτό το μεγάλο ποσοστό. Εδώ έχετε ένα γράφημα όπου το ε, αφορά τον τρόπο με τον οποίο ε, ε, χωρίζονται τα κόμματα όσον αφορά το θέμα του δημοψηφίσματος και 100 είναι η συμφωνία. Και από την άλλη μεριά στο γράφημα βλέπετε με ποιο τρόπο κινητοποιούν τα κόμματα τους, τα μέλη τους. Ε, επάνω αριστερά, στο επάνω αριστερά ε, τετράγωνο βλέπετε ότι ε, έχουμε ας πούμε την υψηλή πυκνότητα των δημοψηφισμάτων όπου οι πολίτες κινητοποιούνται πολύ. Εάν βρίσκεται κανείς λοιπόν σε αυτή την ζώνη το ενδεχόμενο να αποτύχει το δημοψήφισμα πενταπλασιάζεται τα περισσότερα ε, ε, δημοψηφίσματα τα οποία σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση έγιναν για λόγους ε, κομματικούς και έχουμε σε αυτήν την σύγχρονη φάση, δηλαδή μετά από το 2010, μία αυξανόμενη επίπτωση στα πολιτικά και μία αυξανόμενη τάση για αποτυχία. Έχουμε εδώ βέβαια και κάποια στοιχεία στα οποία δεν θα μπούμε σε μεγάλες ε, λεπτομέρειες όσον αφορά δηλαδή την ε, ε, ζήτηση για τέτοια δημοψηφίσματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζήτηση λοιπόν έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Έχουμε για τα κόμματα τα οποία εκπροσωπούνται στην, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η ζήτηση έχει αλλάξει. Αυτά που μέχρι τώρα ήταν μάλλον ε, έτσι ψυχρά ή χαλαρά, χλιαρά απέναντι στα δημοψηφίσματα τώρα έχουν ε, αυξηθεί. Τα κόμματα αυτά δεν είναι τόσο. Έχουμε και άλλα γραφήματα τα οποία περνάω γρήγορα ε, χωρίς να σας τα αναλύω. Αν θέλετε μπορούμε να τα αναλύσουμε μετά ή να σας τα δώσουμε. Σχετικά τώρα με την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2000 ας πούμε, το 2005 και αν το δείτε μέχρι το 2016 ε, είναι μία περίοδος από την οποία, ε, την οποία βλέπουμε σύγκληση των αρνητικών ε, απόψεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ βλέπουμε τις ε, βόρειες χώρες ε, οι οποίες είναι στην Ευρωζώνη και τις βόρειες χώρες που δεν είναι στην Ευρωζώνη όπως ε, η Δανία και μετά έχουμε τις υπόλοιπες χώρες. Βλέπετε ότι η στήριξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση διαφέρει ανάλογα σε ποια γεωγραφική ζώνη βρίσκεται κανείς. Επίσης η στήριξη για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται δηλαδή στην ουσία υπάρχει αυξημένη ζήτηση για πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες θα είναι σε θέση να ε, βοηθήσουν στην υπέρβαση της ε, κρίσης. Το κυριότερο ε, σημείο εδώ, το οποίο δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε, είναι ότι η πολιτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, προχωρά μέσα από πολύ διαφορετικά εθνικά πλαίσια και αυτό στην ουσία δίνει, σχηματίζει τα δημοψηφίσματα και τις διαφορές οι οποίες αντιμετωπίζονται ε, καταλαβαίνετε ότι η εμπειρία άμεσης δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από τις χώρες. Ε, το Βέλγιο δεν έχει τέτοια δημοψήφισμα. Η Ιταλία αντιθέτως έχει πολύ συχνά δημοψηφίσματα. Ένα από αυτά ήταν χτες. Η Ιρλανδία επίσης. Έχουμε λοιπόν διαφορετικές παραδόσεις άμεσης δημοκρατίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τα δημοψηφίσματα γίνονται για διαφορετικούς λόγους στις διαφορετικές ε, ε, χώρες και ρυθμίζονται με διαφορετικά πλαίσια ε, σε, στις χώρες. Στο Λουξεμβούργο, ας πούμε, το πλαίσιο είναι πολύ χαλαρό. Ε, κάτι το οποίο θα αναφέρω αλλά δεν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε είναι ότι έχουν υπάρξει πολλά και ιστάτης ε, ε, σε συγκεκριμένα δημοψηφίσματα από το 2009 και μετά. Θα σας αναφέρω εν συντομία κάποιες, κάποια γενικά συμπεράσματα. Υπάρχει κάτι που ανησυχεί τους ερευνητές ε, δηλαδή ε, αυτή τη δεύτερη σκέψη για τα δημοψηφίσματα, ότι όταν γίνεται δημοψήφισμα δεν ψηφίζουν ακριβώς ε, για το ερώτημα, αλλά υπέρ ή κατά της εθνικής ηγεσία την στιγμή του δημοψηφίσματος. Αυτό είναι προβληματικό. Επίσης βλέπουμε ότι η στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγεί τη συμμετοχή ή όχι και τη στάση που κρατεί κανείς ε, σε ένα ε, δημοψήφισμα. Ε, στην Βόρεια Ευρώπη βλέπουμε ε, πιο εύρο ε, σκεπτιστικές ε, τάσεις και επίσης αυτοί που είναι ευρωσκεπτικιστές έχουν την τάση να μην δίνουν πληροφορίες αφήνοντας την ψήφο τους, την απόφασή τους να την κάνουν τελευταία στιγμή. Ενώ οι φιλοευρωπαίοι είναι αυτοί οι οποίοι δημοσιοποιούν πιο εύκολα την άποψή τους. Αυτό οδηγεί σε κάποια αστάθεια της προετοιμασίας. Επίσης έχουμε διαπιστώσει μια συγκινησιακή βάση ε, των τελευταίων ε, δημοψηφισμάτων όπως ας πούμε για το Fiscal Compact ε, στην Ιρλανδία ή αυτό της Ελλάδος. Τι γίνεται σε αυτήν την σε αυτές τις ε, εκστρατείες ε, ε, είναι ότι η πλευρά του ναι και του όχι τίνουν να φέρονται με άγχος και με θυμό. Επίσης διαπιστώνουμε ότι υπάρχει και μία ανωδική τάση στα λεγόμενα από διαρθρωτικά disintegrative δημοψηφίσματα. Αυτού του είδους ε, τα δημοψηφίσματα ε, αφορούν θέματα πολιτικής ε, και αφορούν κατά κάποιο τρόπο την, τον επαναπατρισμό κάποιων ε, εξουσιών όπως συνέβη ας πούμε στην Ελλάδα το 2015 ή στην ε, Ουγγαρία το 2016. Στην ΔΕ Ελλάδα αγνοήθηκε εντελώς το αποτέλεσμα της, του δημοψηφίσματος. Θα δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφό μου. Στη μελέτη λοιπόν διερευνήσαμε την ε, βιβλιογραφία που είχαμε στη διάθεσή μας σχετικά με το ποιες προτάσεις έχουν διατυπωθεί. Δεν είχαμε αρκετά ευρήματα, παρά το γεγονός ότι είχαμε τέσσερις δεκαετίες ε, δημοψηφισμάτων για ευρωπαϊκά ζητήματα. Όμως, θα μπορούσαμε να δούμε και τις νομικές προκλήσεις μιας συγκεντρωτικής επιβολής, δηλαδή διαδικασία επιπαραβάση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά κάποιων κρατών μελών, επειδή ε, ακριβώς ε, διεξάγουν συγκεκριμένα δημοψηφίσματα που έχουν να κάνουν με αναθεώρηση των συνθήκων. Θα επανέλθω σε αυτό γιατί είναι ένα αρκετά αμφιλεγόμενο θέμα και πολύ λεπτό και πολιτικά φορτισμένο. Δεν είναι ρεαλιστικό πολιτικά, όμως ε, πάρα πολύ έγκριτοι επιστήμονες ε, το έχουν συζητήσει. Εμείς δεν θεωρούμε πως είναι ανέφικτο, ακριβώς διότι οι συνθήκες έχουν μία διατύπωση η οποία προβλέπει κύρωση ή αναθεώρηση των συνθήκων ή διεύρυνση πάντα σύμφωνα με συγκεκριμένες συνταγματικές απαιτήσεις. Και φυσικά γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας υπάρχει το άρθρο 4.2 το οποίο μπορεί, μπορούμε να διτάξουμε σε οποιοδήποτε τέτοιο επιχείρημα για αυτές τις ε, συνθήκων. Θα περάσουμε όμως σε λίγο στη συζήτηση αυτών των θεμάτων. Τώρα, ας περάσουμε λίγο τα τετράγωνα στη δεξιά πλευρά της διαφάνειας, υφιστάμενες προτάσεις δηλαδή στην ε, βιβλιογραφία. Ας δούμε λοιπόν τη βιβλιογραφία κάτω δεξιά, μπορείτε να δείτε. Υπάρχει λοιπόν βιβλιογραφία η οποία διερευνά τις δυνατότητες πανευρωπαϊκού δημοψηφίσματος για, ίδρυτη, για θέματα ίδρυσης Στα μέσα της δεκαετίας του 90 είχαμε τέτοιες προτάσεις, υπήρχε σχολιασμός από μελετητές και πανεπιστημιακούς και μάλιστα πρόσφατα στην Ευρώπη των 28 υπάρχουν ορισμένοι επιστήμονες οι οποίοι προτείνουν διεξαγωγή δημοψηφίσματος για μελλοντικές αναθεωρήσεις των συνθήκων. παρά το γεγονό ότι υπάρχουν ήδη πολύ αυστηροί κανόνες για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, για τα ποσοστά πλειοψηφία κτλ. Εδώ υπάρχει και μία άλλη έρευνα πάνω δεξιά, το πώς μπορούμε δηλαδή να ξεπεράσουμε τη, τα αποτελέσματα μιας ομόφωνης απόφασης. Εδώ υπάρχουν δύο πιθανότητες. Η, η μία πάνω ασύμετρη άμεση δημοκρατία Πώς δηλαδή μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο της ε, διπλής ε, ομοφωνίας επιτρέποντας το κράτος μέλος να χρησιμοποιήσει ε, το δικό του σύνταγμα, να διεξάγει δηλαδή δημοψήφισμα μία χώρα, μία άλλη να μην το κάνει. Η Ιρλανδία ας πούμε δεν μπορεί να ψηφίσει ένα δημοψήφισμα το οποίο θα σταματήσει οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρηση συνθήκων, ακριβώς επειδή η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει καταψηφίσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η άλλη επιλογή είναι άμεση δημοκρατία διπλής πλειοψηφίας. Πολλοί έγκριτοι επιστήμονες του κλάδου προτείνουν κάτι τέτοιο και ο καθηγητής Richard Rose που βρίσκεται εδώ μαζί μας επιχειρηματολογώντας για υπέρ ε, ευρωπαϊκών δημοψηφισμάτων που θα ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια. Και αυτή είναι μια αρκετά αμφιλεγόμενη πρόταση. Τώρα, ε, σε ό,τι αφορά τις δικές μας προτάσεις και συστάσεις. Να πω πολύ σύντομα ότι δεν θα εκπλαγεί κανείς ε, με αυτό που θα πούμε. Πολλά μπορούμε να πούμε για το πώς μπορούμε να αποφύγουμε μεγάλες αναθεωρήσεις συνθήκων. Υπάρχουν ήδη αυστηροί και άκαμπτοι συνταγματικοί κανόνες, όπως και αν ε, τους ε, αναλύσει κανείς, ε, από δικαιώματα βέτο σε εθνικό επίπεδο ή μετά σε υποεθνικό επίπεδο βλέπουμε ότι τέτοιες δυνατότητες βέτο υπάρχουν, όπως με το Βέλγιο για την Συμφωνία ΣΥΤΑ. Υπάρχουν λοιπόν συνταγματικέ προκλήσει, οι οποίες θα εμφανιστούν σε εθνικά δημοψηφίσματα. Εμείς ε, στη μελέτη μας προσπαθήσαμε να χαρτογραφήσουμε αυτές τις προκλήσεις, που έχουν εμφανιστεί τις τελευταίες δεκαετίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά το γεγονός ότι δεν είχαμε αρκετά τέτοια δημοψηφίσματα, αναμένεται να αυξηθεί αυτός ο αριθμός στο μέλλον. Οι κάτω τώρα ε, έχουν επίσης τη δυνατότητα διεξαγωγής δημοψηφίσματος για αναθεώρηση των συνθήκων. Τώρα, για όσους ακολουθήσουν αυτή τη γραμμή, θα μπορούσαμε να προτείνουμε υιοθέτηση πιο τολμηρών ε, επιλογών. Η ομάδα Σπινέλη, για παράδειγμα, έχει προτείνει παρόμοιες ε, ιδέε σχετικά με την άμεση δημοκρατία. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να, να διεξάγουμε ένα δημοψήφισμα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για ε, την αμφισβήτηση υφιστάμενης νομοθεσίας ε, υφιστάμενη νομοθεσία η μικρή κλίμακα άμεση δημοκρατία είναι κάτι πιο εφικτό εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χρησιμοποιήσει τα όπλα που έχει στην συνταγματική της φαρέτρα για να κάνει διάφορες συνταγματικές τροποποιήσεις. Αν δούμε τι γίνεται στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Ιαπωνίας, βλέπουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες για συνταγματικές αλλαγές. Ίσως λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να αναλογιστεί τη δυνατότητα τροποποίησης ή στήριξης διάφορων εκστρατιών για τέτοια δημοψηφίσματα. Επίσης, στη μελέτη προτείνουμε να αμφισβητηθούν κάποιες, ε, κάποια δημοψηφίσματα που μπλοκάρουν περαιτέρω εξελίξεις, περαιτέρω σταγματικές αλλαγές. Ε, όχι βέβαια αναδρομικά, όπως στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά μελλοντικά. Και φυσικά το δημοψήφισμα της Ουγγαρίας είναι ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα στην πρότασή μας. Τώρα, το δημοψήφισμα των κάτω χωρών. Θα μπορούσε να έχει αποφευθεί εάν η Συμφωνία Σύνδεση Ευρωπαϊκή Ένωση και Ουκρανία ήταν κάτι καθαρά διαδικαστικό σε επίπεδο ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια, στο μέλλον, εάν υπάρξει το ενδεχόμενο συνταγματικών αλλαγών, είναι πολύ πιθανό αυτές οι αλλαγές να ε, στεφτούν με επιτυχία δεδομένης της ε, κατάστασης που επικρατεί σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας περάσουμε αμέσως στον καθηγητή Richard Rose. Έχετε το λόγο. Um, Start by. Πρώτα απ' όλα σας... Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ξέρω ότι έχετε ιδιαίτερα βεβαρημένο ε, πρόγραμμα και ξέρουμε πόσο δύσκολα είναι όλα αυτά τα ζητήματα. Κατά δεύτερον θα ήθελα να συμπληρώσω τα όσα υπόθηκαν και να σταθώ στα πολιτικά ζητήματα που ανακύπτουν, γιατί ήδη οι συνάδελφοι ανέφεραν ε, πολύ εμπεριστατωμένα τα νομικά ζητήματα. Το δικό μου σημείο κίνηση είναι ότι όταν αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζω και εγώ γνώμη. Και νομίζω ότι υπήρξε μια διαρθρωτική αλλαγή που τώρα κορυφώνεται ε, με την ε, παραγωγή δημοψηφισμάτων. Ποια είναι η αιτία του προβλήματος. Είναι η αλληλεξάρτηση. Όταν διαμορφώθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν για να σταματήσει ο κίνδυνος ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου και έτσι να ξεκινήσει η γαλλογερμανική φιλία. Έχουν πέρασει πολύ καιρός από τότε, όμως έχουμε οικονομικά ζητήματα παράδειγμα η Ευρωζώνη, προβλήματα εθνικής ασφάλειας όπως είναι η τρομοκρατία στη Γαλλία και μετανάστευση. Και αυτά είναι σημαντικά προβλήματα γιατί ε, ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα, επομένως επηρεάζουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τη νομοθεσία και τις πολιτικές. Πρόκειται για μια αλλαγή λοιπόν στο σημείο εστίασης και έμφασης της πολιτικής. Και όσοι ε, δραστηριοποιούνται στο Ευρωκοινοβούλιο και στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωρίζετε πολύ καλά τα ζητήματα της αλληλεξάρτησης ε, και την ανάγκη εξέβρεσης συμβαστικών λύσεων. Δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο ε, σκέφτονται πολλοί και εδώ εντάσσω και τα μέλη των εθνικών κυβερνήσεων, εθνικών κοινοβουλίων και των εθνικών μέσων ενημέρωση που θεωρούν ακόμα ότι το εθνικό πολιτικό προσκήνιο μπορεί να πάρει τις αποφάσεις για μια χώρα και μόνο αυτό. Στις περισσότερες χώρες ο κόσμος πιστεύει ότι η εθνική κυβέρνηση θα πρέπει ε, να συνομιλεί με άλλες κυβερνήσεις. Δηλαδή δεν θέλουν την απόλυτη απομόνωση, όμως σε τελική ανάλυση οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι και πολίτες μιας χώρας και θεωρούν ότι ως ε, πολίτες ε, μιας χώρας ε, θα πρέπει να αποφασίσουν για μια πολιτική μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης. Δεν πρέπει λοιπόν να κλείσουμε τα μάτια μας προς τον κόσμο. Πρέπει να είμαστε σε θέση να δούμε τι κάνουν οι υπόλοιποι και να πάρουμε μια απόφαση. Η άλλη διαθετική τροποποίηση είναι το κλίμα εμπιστοσύνη για τα γνωστά παραδοσιακά ε, κόμματα και την σύνδεσή τους με το Συμβούλιο. Ξεκίνησε ε, στη Μεγάλη Βρετανία από το 1974 όταν είχαμε η ε, στην Αυστρία στα τέλη της δεκαετίας του 1960 αρχές του 70. που πλέον βλέπουμε ότι έχουν φτάσει την αποδοτικότητα μέχρι το 50% και στην Ιταλία το 1992, στην Ισπανία και τα λοιπά. Έχουμε λοιπόν τα παραδοσιακά κόμματα εξουσίας που αποδέχονται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατανοούν γιατί βρίσκονται εκεί και ε, έχουν ξεπεράσει τυχόν περιορισμού στο παρελθόν. Όμως, οι πρωθυπουργοί και καγκελάροι σήμερα έχουν συγκεκριμένα προβλήματα. Δίλημα του Κολντών, οι υπηρέτες δύο αφεντάδων ήταν το έργο. Αυτό είναι τώρα λοιπόν το δίλημα που αντιμετωπίζουν, γιατί έχουν μία διτή ιδιότητα και πρωθυπουργοί που εκπροσωπούν τη χώρα τους στις Βρυξέλλες, που είναι αρκετά εύκολο αν θέλετε, γιατί είναι ένα πολιτικό έργο Κατά μέσο όρο 49% λάμβαναν ε, ε, οι κυβερνήσεις συνασπισμού. Στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας έχουμε 35% στα μεγάλα κόμματα εξουσίας. Δεν εκπροσωπούν δηλαδή αυτές οι κυβερνήσεις όλους τους πολίτες. Τι σημαίνει λοιπόν με το εθνικό δημοψήφισμα. Περνάμε από την κυβέρνηση συνασπισμού σε ένα συνασπισμό κρατών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και σε ένα συνασπισμό πολυεθνικών πολιτικών ομάδων. Περνάμε λοιπόν σε ένα μεμονωμένο ζήτημα το οποίο αποφασίζεται ακόμα και από το 1% ε, των Ευρωπαίων πολιτών ή στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου 12%, από το 12%. και για να κερδίσει κανείς πρέπει να πάρει πάνω από το 50% των ψήφων. Επομένω, οι περισσότερες κυβερνήσεις θα έχαναν υπό αυτές τις συνθήκες. Από την άλλη, όσοι ψηφίζουν για ένα κόμμα τη αντιπολίτευση ε, ενδέχεται να ψηφίσουν ε, για μια ευρωπαϊκή πολιτική και το κάνουν ε, κάποιε φορέ και συμβαίνει και το αντίθετο. Κάποιοι που έχουν συμφωνήσει με πολιτική στι Βρυξέλλε την καταψηφίζουν μετά στη χώρα του. Έχουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα ότι τα κόμματα εξουσία είναι συνήθω συνασπισμοί διαφορετικών κομμάτων με διαφορετικά συμφέροντα για ζητήματα όπως είναι τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, οι αμβλώσεις Και στα δημοψηφίσματα έχουμε ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί και αυτό είναι το κεντρικό. Τα άλλα τα αφήνουμε κατά μέρο. Αυτό μας οδηγεί σε δημοψηφίσματα, δημοκρατική ψήφο, που κάθε πλευρά μπορεί να κερδίσει. τα ευρωπαϊκά δημοψηφίσματα τελευταία φαίνεται ότι είναι λίγο περιβολικά δημοκρατικά. Ε, συνήθως είναι καλύτερα τα στοιχεία, αλλά όταν φτάνουμε στο 53-47 υπάρχουν προβλήματα. Ήταν καλό αυτό που έγινε στην Αυστρία, αλλά και πάλι έχει το 47% εκεί για το 78% που δεν ήθελε να ψηφίσει ε, τον ε, πρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα εκπροσώπησης. Τι συμβαίνει όταν ε, ένα δημοψήφισμα αντιβαίνει στην ευρωπαϊκή θέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, δυνατότητε επιβολής τη Νομοθεσία εφαρμογής της νομοθεσίας, αλλά είναι κάτι το οποίο θα ήταν αρκετά αντιπαραγωγικό να παρέμβει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με το να ανακηρύξει ας πούμε, παράνομο ένα δημοψήφισμα αν δεν της αρέσει. Και βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, διστάζει να αξιοποιήσει τέτοιες ε, εξουσίες ακύρωση πούμε, των αποτελεσμάτων των δημοψηφισμάτων από τα δικαστήρια. Και αυτό έχει σε με εθνικά ζητήματα και θέματα εφαρμογής. Το ενδιαφέρον σημείο εδώ είναι οι πολυεθνικές αυτές οι υπερεθνικές πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εφόσον εσείς εκπροσωπείτε ως ευρωβουλευτές ε, και έχετε εκλεγεί, δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν έχετε θέση και σχέση με τις εκλογές. Όλοι έχετε εκλεγεί από την εθνική σας εκλογική περιφέρεια. Δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το τι συμβαίνει ε, στην εθνική μας περιφέρεια. Ενώ από διεθνούς άποψης τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ως εκ τούτου... Ένα τρόπος θα ήταν να επιτρέψουμε στις ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες να δαπανούν πόρους σε εθνικά δημοψηφίσματα. Αυτό θα ήταν ε, ίσως ε, μη πρακτικό, θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο και θα ήταν δύσκολο για παράδειγμα για μέλη των εργατικών ε, στην Μεγάλη Βρετανία να πούν ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ένα ευρωπαϊκό δημοψήφισμα στους σοσιαλιστές. θα έπρεπε να διαλέξουμε πολύ με μεγάλη προσοχή, ας πούμε, θα διαλέξουμε τον ε, Μάρτιν Σούλτ ή κάποιον άλλον. Ή τον ε, Κόρμπιν. η πρόταση του Andrew Duff, ας πούμε, που τα οποία θεωρώ αρκετά ενδιαφέρουσα στο Κοινοβούλιο, γιατί καλεί τις πολιτικές ομάδες να προσπαθήσουν να οργανώσουν ή να οργανωθούν σε όλη την Ευρώπη και αυτό συνάδει και με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Η μέση πολιτική ομάδα δεν, είναι, δεν δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρώπη. Επομένω, ε, πρέπει να δούμε σε τι βαθμό είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν ε, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και οι Σοσιαλδημοκράτες. Υπάρχουν λοιπόν ενδιαφέρουσες ε, δυνατότητες και ευκαιρίες που, μπορείτε να διερευνήσετε. Σε ό,τι φορά τώρα ένα δημοψήφισμα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που ανέφερα το 2013, ήταν ότι κατά πρώτον αποφεύγουμε μια εφορία για το ότι μια συμφωνία που κλείνεται στις Βρυξέλλες μπορεί να ευσταθήσει σε εθνικό επίπεδο. Γιατί οποιοδήποτε πρωθυπουργός ή καγκελάριο πρέπει να υπερασπιστεί στην πατρίδα του τα όσα έχουν συμφωνηθεί στις Βρυξέλλες θα έχει πρόβλημα. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχουν και ρήτρε opt-out για τις χώρες εκείνες που δεν θα επιτυχάνουν ε, την διπλή ειδική πλειοψηφία. Αυτή η ρήτρα opt-out είναι διαφοροποιημένη ε, ολοκλήρωση. Αυτό είναι το τελευταίο που θέλω να πω. Γιατί το μέλλον θα είναι η συνασπισμή των προθήμων που αμφισβητούν το δόγμα αλληλεγγύης του 20ου αιώνα. Το σέβομαι, αλλά το αποκαλώ δόγμα του 20ου αιώνα. για τους ε, συνασπισμούς προθήμων υπάρχουν ε, πολλά προηγούμενα. Η ενδιαφέρουσα ιδέα είναι η Σέγγεν, που ξεκίνησε πολύ μικρή και έγινε ένας τεράστιος μαγνήτης. Τώρα απομαγνητίζεται, αν θέλετε να το πω μεταφορικά, όμως ποτέ δεν ήταν ομοιόμορφη. Η Ευρωζώνη ξεκίνησε ως συνασπισμός των προθήμων ε, με έναν τέτοιο λειτουργήσε ως μαγνήτης. Και πάλι κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να απομαγνητιστεί. Αυτές είναι, αυτά είναι παραδείγματα που μας λένε ότι όχι ότι πρέπει να αφήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση Αλλά είναι ενδιαφέρον. Αν ήξεραν για την Ελλάδα όσα ξέρουν σήμερα, ίσως να είχαν κρατήσει διαφορετική στάση. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Επομένω, υπάρχει και μια θεωρία ποδηλάτου. που είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος ε, κοινής, ε, από κοινού κίνησης. Εγώ την, θεωρώ, την, την αποκαλώ θεωρία του μονόκυκλου, γιατί όλοι πηγαίνουν έτσι, ακροβατώντας. Γιατί υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα οικονομικά, πολιτισμικά, πολιτικά, υπάρχουν διαφωνίες, αντιπαραθέσεις μεταξύ χωρών, αλλά και στο εσωτερικό των χωρών. Και για να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα με τις υφιστάμενες συνθήκες είναι πρέπει να ενθαρρύνουμε τους πάντες ε, να συνεργαστούν, να συνομιλήσουν. Και το τελικό μου συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει περισσότερο να επικεντρωθούμε σε συνασπισμούς προθήμων παρά σε μια αλλαγή, διαρθωτική αλλαγή που επιφέρει τροποποιήσεις ε, και στις ε, αλληλεξαρτήσεις από την ε, κοινότητα ΕΚΑΧ και μετά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Το λόγο έχει ο κύριος Φεντερίκο Ντεμελτάλβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θα κάνω την παρουσίασή μου στα ισπανικά. Ε, και θα συνεχίσω στα ισπανικά λοιπόν. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ την Επιτροπή σας που με καλέσατε σε αυτήν την σε αυτήν την εκδήλωση και επίσης να ευχαριστήσω κυρίως και να συγχαρώ τους συγγραφείς ε, της αρχικής παρουσίασης όχι μόνο ε, για την βαθιά τους ανάλυση αλλά και για την συστηματοποιημένη γνώση η οποία μας δίνει τη δυνατότητα με ακρίβεια να μελετήσουμε το θέμα. Εγώ είμαι καθηγητής ε, συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο των Ισουητών της Μαδρίτης και επίσης διδάσκω συγκριτικό συνταγματικό δίκαιο ε, εδώ και 20 χρόνια και εργάζομαι επίσης και για θέματα κυβερνησιμότητας και εκπροσώπησης ε, κομμάτων. Επομένως, κατά την έννοια γνωρίζω το θέμα. Ε, βεβαίως, το κεντρικό ερώτημα δεν είναι μόνο να σχολιάσω αυτή την έκθεση, η οποία είναι εξαίρετη, αλλά και να απαντήσω σε ένα κεντρικό ερώτημα, το οποίο θα πρέπει να απαντήσουμε, δηλαδή, εάν θα πρέπει από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να προωθηθούν τα δημοψηφίσματα και σε επίπεδο κρατών μελών αλλά και σε επίπεδο ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έτσι όπως προτείνεται με ήπιο τρόπο ε, από την έκθεση και αν με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε αυτήν την απομάκρυνση των πολιτών. Κοιτάξτε, είναι μια συζήτηση την οποία ε, ξεκινήσαμε στην Ευρώπη στην αρχή ε, του 20ου ε, αιώνα, τότε δηλαδή που δεν είχαμε ακόμα προσαρμοσμένο πολιτικό μοντέλο έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το τέλος ενός κύκλου. Ε, στην Ευρώπη από το 2004-2005 αναφέρεται ως λύση μέσω μελέτης, να προωθηθεί δηλαδή η λύση του δημοψηφίσματος. Είναι μια ιδέα η οποία θα πρέπει να προωθηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα από το κράτος ε, και την ε, ε, κοινότητα. Ο Αλέξης Δετοκβίλ έλεγε ότι όταν ο διαχωρισμός ανάμεσα στο κράτος και την κοινωνία είναι πάρα πολύ βαθιά, τότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για μια νέα εποχή. Πρέπει οπωσδήποτε να δούμε ότι οι αρχές της ελευθερίας και της αδελφότητας ε, που οδήγησαν μετά από τον δεύτερο ε, παγκόσμιο ε, πρόεδρο, πόλεμο συγγνώμη, ότι πλέον έχουν περάσει σε δεύτερο επίπεδο διότι βλέπουμε δυνάμεις οικονομικές οι οποίες προσπαθούν να μπουν στην δημοκρατική ζωή τα λόμπι τα οποία θέλουν να μπουν στο κοινοβούλιο ενώ απ' έξω μένουν ε, οι κοινωνίες. Δεν ξέρω εάν το ρεφερέντουμ μπορεί να χρησιμεύσει σε αυτόν τον διαχωρισμό. Εγώ όμως ε, θα ήθελα να μελετήσουμε τον, ε, το δημοψήφισμα ως ένα κύριο στοιχείο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας όσο μη τέλεια όσο, ατελούς, ε, όσο ατελής και αν είναι αυτή. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ε, κατά την άποψή μου, είναι εξαιρετικά σημαντική και το λέω, η άμεση δημοκρατία ε, δεν είναι ε, ιδεώδες, δεν υπάρχουν ε, κοινωνίες ελεύθερες όπου ε, υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στους πολιτικούς και τους πολίτες και ούτε εκεί που οι πολίτες θεωρούν ότι πάντα πρέπει να ψάξουν έναν υπεύθυνο ε, στην, ε, παρούμε, ε, στην προκείμενη περίπτωση νομίζω ότι μπορώ να αναφέρω τον William Κώστα, ο οποίος αναφέρεται στην ε, ε, στην ε, κοινωνία των συγχρόνων. Θέλουμε μια δημοκρατία όπου όλοι να συμμετέχουμε και μέσω δημοψηφισμάτων. Δεν είναι τόσο απλό γιατί όλοι ζούμε σε μια περίπλοκη κοινωνία. Ο καθένας μας ασχολείται με τα δικά του θέματα, με τη δουλειά του και επομένως αφήνει τους πολιτικούς να το κάνουν. Τώρα, εάν αν ε, με τη σειρά της ε, η πολιτική ε, μεταφέρει την ευθύνη σε μία, στους πολίτες ή μάλλον σε μία συγκεκριμένη μερίδα των πολιτών αυτό μπορεί να είναι πραγματικά χήμερα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται πάρα πολύ να προχωρήσουν στη δουλειά τους και επομένως δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και πολιτικά όντα. Εγώ δεν θέλω να ε, ε, είμαι αντίθετος προς την κοινωνία των ε, συγχρόνων, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κάτι άλλο ε, είναι να χρησιμοποιηθεί το δημοψήφισμα ε, στα πλαίσια μιας αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Δηλαδή, όχι ε, να χρησιμοποιηθούν με το ζόρι τα δημοψηφίσματα για να προχωρήσει ένα συγκεκριμένο είδος δημοκρατίας, αλλά να χρησιμοποιηθούνται εντός της πρόθεσης της δημοκρατίας. Συνήθως το δημοψηφίσματα τα βλέπουμε εκτός εξαιρουμένες μάλλον της Ελβετίας τα, τα βλέπουμε σε χώρες ε, στις οποίες ε, δεν ε, υπάρχει δυνατότητα για εκλογές. Στην, στην Ελβετία τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ε, στη, επίσης η κοινωνία της ε, Ελβετίας είναι τελείως ε, διαφορετική και καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει τέτοια πολιτική δομή. Απ' την άλλη πλευρά μπορούν να υπάρξουν δημοψηφίσματα για θέματα τα οποία είναι επίγοντα, τα οποία είναι ξαφνικά, τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στην προεκλογική εκστρατεία. Ας πούμε αυτό της Ιταλίας είναι μια καλή μορφή εκπροσωπητική ε, δημοκρατία, όπου ερωτάται ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο σχετίζεται με το Σύνταγμα. Ε, αλλά ε, ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν και τοπικά δημοψηφίσματα τα οποία είναι τελείως διαφορετικά. Σε αυτή την περίπτωση τα δημοψηφίσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν την οδό προς την δημοκρατία. Κοιτάξτε, τα, είναι γεγονός επίσης και αυτό αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι τα δημοψηφίσματα απομακρύνουν ακόμα περισσότερο τον κόσμο από την ε, πολιτική. Δηλαδή μέσω της κριτικής ε, ε, ενισχύουν την, την απομάκρυνση του πολίτη ενώ υποτίθεται ότι έχουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Μειώνουν επίσης τον πλουραλισμό γιατί η απάντηση είναι ναι ή όχι. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο, δεν υπάρχει γκρίζο και επομένως υπάρχει μόνο νικητής και ηττημένος. Αλλά ξέρετε ότι στην πολιτική δεν είναι έτσι. Και Επομένως ε, η κοινωνία είναι πολύ πιο περίπλοκη και δεν είναι δυνατόν ε, να μπαίνουμε σε μια διαδικασία δημοψηφίσματος σε μια τέτοια σύγχρονη κοινωνία η οποία χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο φάσμα και τελικά να πρέπει να απαντήσουμε με ένα ναι ή με ένα όχι. Από την ε, άλλη πλευρά όταν στα δημοψηφίσματα βλέπουμε ότι παίζουν ρόλο τα συναισθήματα και οι συγκινήσεις είναι πρόβλημα γιατί η πολιτική πρέπει να γίνεται με τη λογική. Ε, ε, ε, επίσης, Επίσης στην Ευρώπη πρέπει να πούμε ότι γίνεται μια προσπάθεια να να δημιουργηθεί μια νέα ε, διαδικασία η οποία υπάρχει στη Βόρεια Αμερική αλλά όχι σε εμά. Ε, αυτήν την έννοια ας πούμε του ε, επιτηρητή της, της και καταλαβαίνετε ένας λαός δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει με διαφορετικό τρόπο στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία. Όντως έχουμε διαπιστώσει ότι μπορεί να δημιουργηθεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μέσο για να ε, μειωθούν ε, οι εντάσεις. Ε, μπορούμε επίσης να το χρησιμοποιήσουμε για να προχωρήσουμε σε καταστάσεις, σε μοντέλα διαφορετικά. Γιατί λένε είμαστε σε κρίση. Αλλά εγώ θυμάμαι ότι μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτό το λογικό αντιπροσωπευτικό μοντέλο έτσι όπως το αναπτύξαμε και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μοντέλο ακριβώς έτσι ώστε να αποφευχθεί το τι, αυτό που συμβαίνει αλλά και έτσι ώστε να βελτιωθεί, να λυθεί καλύτερα αυτό που συμβαίνει. Αλλά εδώ φτάνουμε σε ένα παράλογο. Ε, ε, ε ακριβώς αυτό που επιτυχάνουμε προσπαθούμε να το τροποποιήσουμε. Ε, υπάρχει και ένας Ισπανός, ο Ντανιέλ ε, ο οποίος συνήθως γράφει στα Ισπανικά, αλλά σε ένα επιστημονικό άρθρο που ονομάζεται «Η δημοκρατική απογοήτευση» λέει ότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, αντιπροσωπικη δημοκρατια μιλάει για δημοκρατία αλλά μιλάει για την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, είναι ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δημιουργεί διαρκώς την εξαίρεση κυρίως όταν λειτουργεί σωστά. Διότι ε, ε, τα, ε, διότι αντίθετα από τα νέα μοντέλα, δημοκρατικά ή μη δημοκρατικά, δεν το κάνουν. Ε, στην ουσία δηλαδή λέει ότι οποιαδήποτε, οποιαδήποτε μοντέλο λογικής δημοκρατίας οδηγεί στην απογοήτευση. Και ακριβώς αυτή η απομάκρυνση, η απογοήτευση από την δημοκρατία είναι ένα φυσικό φαινόμενο αναμενόμενο γιατί οδηγώντας τον λαό προς τα ιδεώδη της δημοκρατίας, πάντα ελπίζουμε περισσότερα, προσδοκούμε περισσότερα ε, και επομένως και αυτοί που περιμέναν τα περισσότερα και αυτοί που περιμέναν τα λιγότερα στην ουσία, ε, στην ουσία βλέπουν τις προσδοκίες τους να διαψεύδονται. Εγώ ως ένας απλός καθηγητής πραγματικού δικαίου λέω ότι και σε τοπικό ε, επίπεδο όντως μπορούν να δημιουργούνται, να οργανώνονται τέτοιου είδους δημοψηφίσματα αλλά κυρίως λέω ότι θα πρέπει να διοργανώνονται ακριβώ για να αποφεύγονται καταστάσεις σαν αυτή ε, που συζητούμε τώρα. Ε, ας ε, θυμηθείτε ε, τι έκανε ο Καρέλ ο Χάνς Καρέντε Μαλμπέργ ή ο Χάνς Κέλσεν στο, στην αρχή του 20ου αιώνα που έλεγαν ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε τον δεσμό ανάμεσα στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ανάμεσα στον εκπρόσωπο και τον εκλογέα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να εκπαιδεύσουμε πλέον τις νέες γενιές στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία ε, και να πιστέψουμε ότι οι νέες γενιές δεν θα έχουν τόσο μεγάλη προσκόλληση και αγάπη προς την δημοκρατία όσο είχαμε εμείς οι παλαιότερες γενιές. Ε, πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε ε, να εισάγουμε και την ιδέα του δημοψηφίσματος που ένα χρόνο πριν έλεγε κάποιος ότι θα μπορούσε να είναι μια καλή δομή αλλά που εν πάση περιπτώσει είναι μια δομή εξαιρετικά επικίνδυνη και το τονίζω επικίνδυνη επικίνδυνη. Αυτό ήθελα να πω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά τους ε, συγγραφείς ε, για την, τις για την ανάλυση, αλλά και για, την, ε, και για όλα τα στοιχεία τα οποία επιτρέπουν μία σωστή διάγνωση. Ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε στη συζήτηση τώρα. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο Γιώργη Σόπφλιν. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εκ μέρου του ΕΛΚ θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να πω πως ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ακούσαμε. Ε, ήμουν και εν μέρη υπεύθυνο για αυτήν την κουβέντα, γιατί είχα προτείνει την ακρόαση για αυτό το θέμα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε διάφορα ζητήματα. Καταρχάς, νομίζω πως ε, αυτά που είπε ο Μάριο Μέντες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ε, ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Ήμουν ο ίδιο εισηγητή για τη σχετική έκθεση και έχω τι δικέ μου προσωπικέ απόψει. Εγώ δεν θεωρώ πω ε, αυτή η πρωτοβουλία είναι ένα ε, μέσο άμεση δημοκρατία, διότι απαιτούνται ένα εκατομμύριο υπογραφέ αντί για 500.000. Υπάρχει δηλαδή, είναι δηλαδή πολύ ψηλά ο πύχης. Μετά, αν δούμε το άρθρο 11, θα παρατηρήσουμε ότι καλή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι αναφέρει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια μπορεί να αρνηθεί την πρόσκληση αυτή. Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Δεν είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Λυπάμαι που το λέω. Αλλά αν δούμε τα στατιστικά στοιχεία, θα δούμε ότι υπάρχουν 58 μέχρι τώρα πρωτοβουλίες με 100% ποσοστό αποτυχίας χρησιμοποιήσαμε όλα τα μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας, αλλά αποτύχαμε παταγωδός. Υπάρχει λοιπόν ένα σημαντικό πρόβλημα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την αποτυχία της πρωτοβουλίας των πολιτών. Δεν θα επεκταθώ σήμερα. Όμως δεν ξέρω εάν, εάν αυτό που είπατε αποτελεί κριτήριο για την άμεση δημοκρατία. Είναι περίπτωση ιδιάζουσα αλλά ξέρω πως υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες ε, είναι αποτελεσματικές. Αν όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνηθεί να αντιδράσει δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έχουν γίνει διάφορες τέτοιες πρωτοβουλίες, έχουν υπάρξει κινήσεις χωρίς όμως αποτέλεσμα. Αλλά κάποιος από εσάς, ε, δεν θυμάμαι ποιος, ανέφερε το δημοψήφισμα στην Ουγγαρία. Ε, καταλαβαίνω τι λέτε, ως ας μην παραμελούμε την εγχώρια διάσταση του δημοψηφίσματος στην Ουγγαρία. Είχε να κάνει πολύ με την εγχώρια πολιτική και χρησιμοποιήθηκε ως αφορμή για να κινητοποιηθεί ο πληθυσμός της χώρας και αυτή η κινητοποίηση πέτυχε και μάλιστα η κυβέρνηση του Φίντες ήταν αυτή που ανέβασε το όριο στο 50% στο δημοψήφισμα. Από την άλλη όμως ήταν και η πρώτη φορά που η κυβέρνηση του Φιντές, εντάξει το λέω γιατί ανήκω και εγώ σε αυτό το κόμμα, αλλά ήταν η πρώτη φορά που η κυβέρνηση του Φιντές κατάφερε να φέρει 3,3 εκατομμύρια Ούγγρους στις κάλπες. Ε, τώρα, εάν παρατηρήθηκε, αν εσείς λέτε πως υπήρξε κατάχρηση η κακή χρήση του δημοψηφίσματος, αυτό είναι η άποψή σας. Όμως από την άλλη υπήρξε αυτή η κινητοποίηση και δεν μπορείτε να λέτε πως ε, το σωστό θα ήταν να, ε, πει, να πούν στους πολίτες όχι μην ψηφίσετε. Οι πολίτες ψήφισαν και υπάρχουν επιπτώσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής στα κράτη-μέλη. Τώρα, να πω και κάτι άλλο. Όταν γίνεται δημοψήφισμα για ευρωπαϊκά ή κοινοτικά ζητήματα, συνήθως γίνεται για να αντιδράσει στους τεχνοκράτες, την τεχνοκρατική προσέγγιση που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτός είναι, αυτή είναι και η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πάρα πολλούς πολίτες. Ε, δυστυχώς, πρέπει να φύγω πολύ σύντομα, γιατί έχω μια ομάδα επισκεπτών και θα πρέπει να τους εξηγήσω τι ακριβώς κάνουμε εμείς εδώ αλλά να σας πω ότι πολύ συχνά όταν έχω τέτοιες ομάδες ε, με κοιτάζουν με βλέμμα γελάδας. Δεν καταλαβαίνουν τι τους λέω. Δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται ούτε σε αυτό το κτίριο, ούτε στις Βρυξέλλες γενικότερα. Ε, κάτι άλλο που ήθελα να πω. Αφορά τα δημοψηφίσματα και το, το Δήμο της Ευρώπης, το λαό της Ευρώπης. Νομίζω πως δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, νομίζω πως ε, αυτές οι εποχές έχουν παρέλθει και το γαλλικό και το ολλανδικό δημοψήφισμα το 2005 έκλεισαν αυτή την πόρτα, είπαν όχι. Αυτό που χρειάζεται είναι να ενισχυθεί η φωνή των πολιτών στις, ε, στα κρατημέλη και ακριβώς μέσω ε, των εθνικών ε, ψηφοφοριών. Τέλος. Θα ήθελα να πω κάτι στον ε, καθηγητή Ροούς και να τον συγχαρώ παρεπτόντος. Να πω ότι δεν ξέρω εάν έχουν αλλάξει ριζικά τα πράγματα από, τις, από την εποχή ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά εγώ πιστεύω πως ο κύριος σκοπός είναι η επίλυση διαφορών και πιστεύω ότι εδώ ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια σχετική επιτυχία παρά το γεγονό, ε, εντάξει σίγουρα δεν έχει ξαναγίνει πόλεμος Γαλλίας-Γερμανίας αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Ας σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο μου είναι αρκετά ε, κοντινό. Πρόσφατα ο Τρέν Μπασέσκου, πρώην Πρωθυπουργός της Ρουμανίας, είπε ότι η Ρουμανία πρέπει να έχει σύνορα ε, στον ποταμό Τίσα να φτάνουν μέχρι εκεί τα σύνορα και ο ποταμός αυτός φτάνει 50 χιλιόμετρα μέσα στην Ουγγαρία. Υπάρχει δηλαδή μια αμφισβήτηση ε, από, που, των σύνορων από το 1916. Αυτό σίγουρα είναι ένα ε, πρόβλημα. Υπάρχει δηλαδή μια ε, ξεκάθαρη αξίωση εδαφική τη Ρουμανία σε ουγγρικό έδαφο. Όμω κανεί δεν ανησύχησε στην Ουγγαρία γιατί γνωρίζουν όλοι ότι δεν, δεν ήταν σοβαρή αυτή η αξίωση διότι είναι και οι δύο χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα ήταν προεκλογικό τέχνασμα της... Ε, ε, που χρησιμοποιήθηκε στη Ρουμανία για να κερδίσουν τις εκλογές, όμως δεν ίδρωσε και ταυτή Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μπρέσο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ιταλικά. Α, βάλτε λοιπόν τα ακουστικά σας. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω θερμότατα τους προσκεκλημένους μας. Ήταν πολύ ενημερωτικές οι παρουσιάσεις σας για τα διαφορετικά δημοψηφίσματα, τους διαφορετικούς τύπους δημοψηφίσματος στις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πραγματικά υπάρχει μια τάση που την παρατηρούμε όλοι. Αυτό είπε και ο συνάδελφος εξάλλου, το είπατε κι εσείς, ότι δηλαδή χρησιμοποιείται το δημοψήφισμα για εθνικούς σκοπούς. Έτσι ώστε δηλαδή να δώσουν στους πολίτες μία διαφορετική επιλογή. η οποία θα αλλάξει την μέχρι τώρα σχέση τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ συχνά βέβαια βλέπουμε ότι οι ερωτήσεις στα δημοψηφίσματα είναι έτσι διατυπωμένες ώστε να προκαλούν σύγχυση. Πολλές φορές μάλιστα δεν είναι και σωστή η διατύπωση, δεν υπάρχει συμφωνία με τις συνθήκες. Εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα το Βρετανικό δημοψήφισμα που είχε να κάνει με αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένο μια κυβέρνηση να συμβουλεύεται τους ε, πολίτες της για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις που ένα δημοψήφισμα δεν είναι σωστό, διότι ο πολίτης δεν καταλαβαίνει την ερώτηση. Προσπαθεί δηλαδή μια χώρα να αλλάξει τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά το γεγονός ότι έχει συμφωνήσει για αυτή τη σχέση μέσω υπογραφής συνθήκων. Εσείς τι άποψη έχετε για αυτές τις περιπτώσεις δημοψηφισμάτων. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω την άποψή σα και εντάξει αν όχι τη λύση στο πρόβλημα γιατί σίγουρα είναι μεγάλο κάποιες προτάσεις, τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στα πλαίσια των συνθήκων, τι μας επιτρέπεται. Υπάρχει δυνατότητα να απαγορευτούν τέτοιου τύπου δημοψηφίσματα. Υπάρχει κάποια σαφής διατύπωση σχετικά με το τι μπορεί, τι ερώτηση μπορεί να τίθεται σε ένα δημοψήφισμα, αν επιτρέπεται να ερωτάτε η άποψη των πολιτών για τόσο σοβαρά ζητήματα όπως παραμονή ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα αντιδρούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Διότι σίγουρα όταν κάποιος υπογράφει μία σύμβαση δεν μπορεί να χωρί από αυτή τη σύμβαση έτσι απλά. Ας πούμε λοιπόν ότι ένα κράτος ε, επιθυμεί να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι δυνατότητες έχει. Υπάρχει μια σύμβαση η οποία έχει επικυρωθεί, δεν γίνεται κάτι και πώς λοιπόν ένα κράτος που επιθυμεί να αποχωρήσει μπορεί να το καταφέρει μέσω δημοψηφίσματος, μέσω κάποιας άλλης ε, δυνατότητας. Εσείς τι ε, άποψη έχετε. Μπορεί να δοθεί κάποια διαφορετική ερμηνεία σε συγκεκριμένες διατάξεις των ε, συνθήκων έτσι ώστε να παγουρευτούν τέτοιου τύπου ε, πολιτικές σκοπιμότητες στα δημοψηφίσματα. Δεν είναι αστείο το θέμα. Δεν μπορούμε ε, να το αντιμετωπίζουμε με ευθυμία. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Εάν κάποιος θέλει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε πρέπει να τηρούνται ορισμένοι κανόνες και όχι να χρησιμοποιούνται ε, πολιτικές σκοπιμότητες για να αλλάξουν οι συνθήκες ε, προς ε, όφελος κάποιου κράτους. Ευχαριστώ πολύ πούμε παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Περισσότερο παρατηρήσεις, όχι τόσο ερωτήσει για τα όσα υπόθηκαν από τους ομιλητέ μας σήμερα. Είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχω εκλεγεί από μια εκλογική περιφέρεια στη Γαλλία. Νομίζω ότι η χώρα μου ήταν από τις πρώτες ε, που ξεκίνησε τους τελευταίους δύο αιώνες ε, αυτή την πολιτική των δημοψηφισμάτων. Όμως κάθε φορά ε, αποτελούσε μία εκλογική παρέκκληση. Αυτό συνέβη κατά την ε, περίοδο του Ναπολέοντος του Πρώτου και του Τρίτου που ε, αξιοποίησαν αυτό το δημοψήφισμα για εκλογικούς σκοπούς και πάντα ήμασταν πολύ φιδωλοί ε, στην χρήση ε, των δημοψηφισμάτων στην σύγχρονη εποχή. Υπενθυμίζω ότι το Γαλλικό Σύνταγμα προβλέπει τη δυνατότητα εξαγωγής δημοψηφίσματος σε μια πλειάδα άρθρων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό ποτέ δεν είναι υποχρεωτικό το δημοψήφισμα ε, για τις αρχές. Εκτός από μία και μόνη περίπτωση που αφορά ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Μπορείτε να αλλάξετε το σύνταγμα, το γαλλικό σύνταγμα, έχει τροποποιηθεί πολλές φορές ε, με ειδική ε, κοινοβουλευτική πλειοψηφία των δύο σωμάτων. Μπορείτε να την τροποποιήσετε όσο θέλετε λοιπόν το γαλλικό σύνταγμα και εκεί δεν χρειάζεται να κάνετε το δημοψήφισμα ε, μόνο μία περίπτωση υποχρεωτικής εξαγωγής των τη υπάρχει από το 2007. Δεν έχουμε αξιοποιήσει λοιπόν για ευρωπαϊκό ζήτημα αφορά την ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας χώρας που δεν ανήκει στον κατάλογο της ε, Διακυβερνητικής Συμφωνίας του 2004. Επομένως πρόκειται για μια προφορική γραπτή παράκαμψη για να μην μπούμε Τουρκία ουσιαστικά. Η μοναδική χώρα που θα μας ενδιέφερε σε μια πιθανή μελλοντική ε, διεύρυνση δεν θα ήταν ε, η περίπτωση μιας βαλκανικής χώρας, θα αφορούσε την περίπτωση της Τουρκίας. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν το δημοψήφισμα θα ήταν υποχρεωτικό. Υπάρχει δικαίωμα άρνηση κυρίας του γαλλικού λαού για το σύνολο των αποφάσεων των υπολείπων κυβερνήσεων ή των ε, γνωμοδοτικών συμβουλευτικών δημοψηφισμάτων όπως αυτό στην Ολλανδία. Υπενθυμίζω ότι στην Γαλλία μπορούμε να κάνουμε δημοψηφίσματα. Αυτό συνέβη και το 2005 για την ε, ε, υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Έγινε για εσωτερικούς πολιτικούς ε, λόγους το δημοψήφισμα. Χάθηκε. Μετά είχαμε προεδρικές εκλογές δύο χρόνια αργότερα που ουσιαστικά ενέκριναν το αντίθετο του δημοψηφίσματος και έτσι υιοθετήθηκε. Εγώ είμαι ένθερμος υποστηρικτής, ξέρετε κύριε Μολτάβο, της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Προσωπικά είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικό ό,τι αφορά την χρήση ε, των δημοψηφισμάτων, επειδή υπάρχει αυτός ο πολιτικός χαρακτήρας και ε, ε, μη αναστρέψιμος χαρακτήρας του κάθε δημοψηφίσματος, ακόμα και όταν ε, κερδίζει κανείς μία από τις δύο επιλογές για λίγο. Επομένω, όταν πρόκειται για, μία, για ένα νόμο που μπορεί ακόμα και να χαίρει τη πλειοψηφία των τριών πέμπτων, μπορεί να τύχει ο νομοθέτης ε, να κάνει λάθος, να τροποποιηθεί σε 10, 20, 50 χρόνια. Και γενικά ε, εγκρίνουμε, θεωρούμε ότι έχει εγκριθεί όταν πρόκειται για δημοψήφισμα ή μπορεί να έχει ταχύτατα μη αναστρέψιμες επιπτώσεις. Ε, η απόφαση να διεξαχθεί δημοψήφισμα στην Αγγλία, εγώ δεν είμαι ε, υποτελής ε, της αυτού μεγαλειότητος, όμως αυτή η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο μιας ε, εκλογικής αναμέτρησης που ε, θεωρεί, θεωρεί το περίπλοκη και γι' αυτό αξιοποιήθηκε αυτό το μέσο. ακολουθώντας μία απόφαση που είχε ληφθεί ε, μέσω δημοψηφίσματος πριν από 30 χρόνια για την ένταξη. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο μη αναστρέψιμο ε, χαρακτήρα ενώ πάντα πρόκειται για ένα πολιτικό ζήτημα, πολιτικών σκοπιμοτήτων. Πάντα έτσι ξεκινάει. Εάν πρόκειται τώρα για δημοψηφίσματα κατόπιν πρωτοβουλία πολιτών και πάλι είμαι αντίθετο, γιατί πρόκειται για ζητήματα που θέτουμε ε, σε δημοψήφισμα γιατί υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια άτομα που απαιτούν να τεθεί σε δημοψήφισμα το ερώτημα αυτό. Και κάθε φορά η εμπειρία μας δείχνει ότι όταν τίθεται σε δημοψήφισμα το ερώτημα ε, τα ποσοστά συμμετοχή είναι πολύ χαμηλά. Τα ποσοστά συμμετοχή όμως εν γέννη δεν ε, λαμβάνονται υπόψη για την αναγωγή συμπερασμάτων από ένα δημοψήφισμα. Και έτσι έχουμε τελικά μία απόφαση αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ε, αντίθεσης ε, ε, κατάργησης μίας συνθήκη από ένα δημοψήφισμα που μπορεί να έχει αποτέλεσμα τελικά 52% αλλά με πολύ χαμηλά ποσοστά συμμετοχής γιατί δεν είναι υποχρεωτική ψήφος. Επομένω, είμαι αρκετά επιφυλακτικό και απέναντι σε αυτά τα δημοψηφίσματα πρωτοβουλία πολιτών που μπορούν τελικά να οδηγήσουν ε, σε μια τυραννία των μειονοτήτων όταν ε, ξεπερνάμε τη λογική. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε για ένα δημοψήφισμα. Αν κατάλαβα καλά, αυτό σημαίνει ότι διοργανώνουμε ένα δημοψήφισμα σε ε, ευρωπαϊκό ζήτημα, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, όπου όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες ψηφίζουν την ίδια ημέρα. Ήδη το να συμφωνήσουμε για την ημέρα θα είναι αρκετά δύσκολο. Άλλοι ψηφίζουν Κυριακή, άλλοι Δευτέρα, Τρίτη. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε λοιπόν από πριν. Επομένω θα πρέπει να ψηφίσουμε την ίδια ημέρα για ένα ζήτημα. Και να λέμε ψηφίζουν σε Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ελετονία κτλ. και έχουν την ίδια βαρύτητα. Μετά, λαμβάνουμε υπόψη το αποτέλεσμα. Ε, ένα πλειοψηφικό αποτέλεσμα, ε, στο 60%. Αλλά στη μία ή την άλλη χώρα έχουμε το αντίστροφο αποτέλεσμα. Κατά χώρα φαντάζομαι θα γίνει η την αλλη χωρα εχουμε το αντιστροφο αποτελεσμα κατα χωρα φανταζομαι θα γινει κατά μέτρηση των ψήφων. Φανταστείτε λοιπόν Έχουμε ένα ζήτημα το οποίο δεν λαμβάνει την πλειοψηφία ε, στη Γαλλία, αλλά λαμβάνει την πλειοψηφία στις υπόλοιπε χώρες τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Όταν εδώ μιλούμε για την επικουρικότητα συνεχώ. για την τήρηση και τον σεβασμό προς την αυτοδιάθεση ε, και την εθνική κυριαρχία των ε, χωρών. Απευθείας βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο, πολιτικό και θεσμικό αδιέξοδο, το οποίο θεωρητικά οδηγεί στην ε, τελική ε, ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού φεντεραλισμού, όμω στην πράξη πρόκειται για απόλυτη αποτυχία. Στη Γαλλία, ε, μπορώ να σα πω πολύ συγκεκριμένα, ποτέ δεν απαντούμε ε, στο ερώτημα που μα τίθεται. Ποτέ. Και αυτό είναι το ζήτημα που χάνουμε τελικά. Πρόκειται πάντα για μια εκλογική εκστρατεία άλλες ε, σκέψεις, ιστερόβουλες κινήσεις για τις επερχόμενες εκλογές που γίνονται κατά μέσο όρο κάθε 16 με 18 μήνες. Ακόμα και αν ένα ζήτημα λοιπόν ενδιαφέρει τους πάντες, καταψηφίζουμε για να διώξουμε την κυβέρνηση που έχει προτείνει ένα ζήτημα. Ακόμα και εκείνη που θα ήταν υπέρ της, αντι, της αντιπολίτευσης θα ψήφιζαν αντίθετα. Ξέρετε τώρα πώς πάει αυτό, όπως έγινε και στην Ιταλία. Επί της αρχής λοιπόν, ναι, όπως όλοι ε, φαντασιώνονται την ελληνική δημοκρατία, την αγορά και ούτω καθεξής. Όμως βέβαια ποιοι ήταν αυτοί που ψήφιζαν, οι ε, διοκτήτες των σκλάβων. Ούτε οι σκλάβοι ούτε οι γυναίκες είχαν δικαίωμα ψήφου. Επομένω πρέπει ε, να την εξετάζουμε με κάποια περίσκεψη και την αρχαία ελληνική δημοκρατία. Όμω και τώρα βλέπουμε λοιπόν ότι πέραν των φαντασιώσεων είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά συμμετοχή και πολύ σημαντικέ αδυναμίε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζέιμ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και ε, κύριοι ομιλητέ, σα ευχαριστώ και του τέσσερι για τι παρουσιάσει σα. Ντάιαν Τζέιμ ονομάζομαι, είμαι ευρωβουλευτή από, από το Ηνωμένο Βασίλειο και ήμουν μέλο του UKIP μέχρι πριν από μερικέ ημέρε. Επομένω, καταλαβαίνετε ότι θα θέσω ερωτήματα, υπό το πλαίσιο όμως της ενεργού μου συμμετοχής ε, στην εκστρατεία για την αποχώρησή μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινώ με κάποιες παρατηρήσεις με βάση σχόλια που κάνατε, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να τα θέσουμε επιτάπητος. Πρώτον, οι ευρωσκεπτικιστές λένε ότι είπατε, χρειάζονται λιγότερες πληροφορίες και στοιχεία. Θα σας υπενθυμίζω ότι είχαμε τρεις πρωθυπουργού από το 1997 και μετά, Blair, Brown και Cameron το 2010, που και οι τρεις ε, απαρνήθηκαν την άμεση δημοκρατία αναφέροντας σε μανιφέστο ότι θα μπορούσαν ε, και μάλιστα δεσμεύτηκαν να δώσουν ε, και να διοργανώσουν δημοψήφισμα και μετά το αποκήρυξαν. Επομένω, είχαμε μια αυξημένη ανάγκη και ε, διατήρηση των πληροφοριών αυτών. Δεύτερον, είπατε ότι κάποια δημοψηφίσματα οδηγούν σε ε, ανακίνηση των παθών, ε, του θυμού και της ε, αγωνίας. Όμως βλέπουμε ότι τα δημοψηφίσματα σε πολλές περιπτώσεις οδηγούν αυτή την πολιτική, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο πρόκειται για τα μέσα ενημέρωσης ή για την πολιτική σκηνή που ασχολείται με όλα αυτά. Φέτος η κυρία Χάμς, ε, επικεφαλής των Πρασίνων, είπαν, είπε σε ομιλία της, ότι θέλει να καταργήσει ε, τα εθνικά δημοψηφίσματα γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και παραθέτω. Και ανέφερε ότι αυτός ο κίνδυνος ε, επιμόλυνση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ ψηλός και δεν μπορούμε να το δεχθούμε αυτό το ενδεχόμενο. Επομένω, τα ερωτήματά μου προς εσά, βάσει και των όσων ανέφερε η κυρία Μπρέσο. Εσείς θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ακολουθήσει αυτή την οδό που ανέφερε η κυρία Χάμς. Θεωρείτε λοιπόν ότι ε, η σύσταση που θα κάνετε θα είναι αυτή. Γιατί όταν δημοσιοποιηθεί αυτό, σας διαβεβαιώ ότι θα υπάρχουν έντονες ε, αντιδράσεις σε όλη την Ευρώπη. Και χαριτολογώντας η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι αυτή που θα αποφασίσει να καταργήσει τα εθνικά δημοψηφίσματα ή θα συμπεριληφθούν και τα εθνικά κοινοβούλια στη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κανεί άλλο ε, το λόγο. Να θέσω και εγώ ορισμένα ερωτήματα λοιπόν, γιατί δεν έχουμε χρόνο, μόνο 10 λεπτά. Αναλύσατε συστηματικά πολλά ε, δημοψηφίσματα, καμιά 70 περίπου. Να σας ρωτήσω το εξής. Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής τυπολογίας, μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα δημοψηφίσματα τα οποία ήταν πραγματικά ε, μια, ε, μια πρωτοβουλία των πολιτών και δεν ξεκίνησαν από κομματικά συμφέροντα. Επίσης, εδώ και 60 χρόνια ε, έχουμε την εθνική ε, δημοκρατία την οποία εδώ και 60 χρόνια προσπαθούμε να ε, περάσουμε σε ένα πιο διεθνές έτσι, υπερεθνικό επίπεδο. Ίσως καταφέραμε να κάνουμε ένα τέτοιο βήμα προς την υπερεθνική δημοκρατία, αλλά βλέποντας φυγομετρήσεις της κοινή γνώμης και βλέπει κανείς ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, στην ουσία δεν ε, εκπροσωπεί Πραγματικά, δεν αισθάνεται ο κόσμος ότι εκπροσωπείται πραγματικά από το Κοινοβούλιο και από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύετε ότι το γεγονός ότι δεν ταυτίζονται ακόμα οι πολίτες με την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία ε, αποτελεί και έναν από τα στοιχεία τα οποία οθούν ε, στην απέτηση δημοψηφισμάτων επί ευρωπαϊκών θεμάτων. Ο Τζορ Σέπλινγκ τα είπε και προηγουμένως σχετικά με τις ε, πρωτοβουλίες των πολιτών. Βλέπουμε ότι ε, και μετά την συνθήκη της Λισαβόνας ε, δεν έχουμε αρκετό χώρο για την συμμετοχική δημοκρατία έτσι ώστε να συμμετέχουν οι πολίτες στις αποφάσεις που λαμβάνονται. Από αυτήν την άποψη έχει αυξηθεί η όρεξη των πολιτών να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης απόφασης ε, και κατά κάποιο τρόπο με αυτή την έννοια είναι λίγο απαρχαιωμένες οι συνθήκες μας. Συμφωνείτε λοιπόν μαζί μου ότι από αυτή την άποψη οι ευρωπαϊκές συνθήκες ε, δεν είναι και πολύ επίκαιρες ε, τρίτον. Ε, επίσης ε, έχουμε διάφορα δημοψηφίσματα με το ίδιο θέμα. σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορείτε να μας το σχολιάσετε. Ναι, θα ξεκινήσω εγώ γιατί πολλά είναι τα ζητήματα τα οποία αφορούν και συνταγματικά ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες ε, και τα δημοψηφίσματα. Πολύ σύντομα, γιατί ξέρω ότι ο Φερνάντο θέλει να απαντήσει μετά, για το θέμα του, ε, της πρωτοβουλίας των πολιτών. Είναι ένα είδος... Ε, άμεσης δημοκρατίας θα πει περισσότερο Φερνάνδο γι' αυτό και πιστεύω ότι δεν είναι καλό να λέμε ότι είναι απόλυτη η αποτυχία ε, ε, το γεγονός του ενός εκατομμυρίου ε, των υπογραφών νομίζω ότι είναι ήδη κάτι θετικό. Μπορεί να θεωρηθεί ένα καλό στοιχείο και υπήρξαν ε, και ακροάσεις ε, σχετικές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις οποίες εγώ θα μπορούσα να ονομάσω επιτυχημένες, σχετικά με το θέμα της Ουγγαρίας και να απαντήσω εν μέρη με τον τρόπο αυτό στην ερώτηση σχετικά με την ε, απαγόρευση, κατάργηση των δημοψηφισμάτων. Το θέμα του δημοψηφίσματος της Ουγγαρίας νομίζω ότι αποτελεί ε, κατάφορη κατάχρηση ε, των ε, κειμένων των συνθήκων. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό. γιατί ελήφθη απόφαση για δημοψήφισμα ε, για θέμα δεσμευτικό ευρωπαϊκού θέματος ενώ σχετικό άρθρο αναφέρει ότι δεν είναι δυνατόν να ληφθούν, να γίνουν δημοψηφίσματα σε σχέση με θέματα τα οποία έχουν ήδη αποφασιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, και νομίζω ότι ανέτος ναι, μπορούμε να πούμε ότι ε, η από συνταγματική άποψη δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουν τέτοιου είδους δημοψηφίσματα. Για το θέμα των ε, ευρωπαϊκών δημοψηφισμάτων φαντάζομαι ότι ο πρόεδρος, ε, ο κύριος Ρόουζ δεν θέλει να παρέμβει ε, και ο εκδεξιών μου, ο Φερνάντο. Σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Μπρέσο, ναι, υπάρχουν, υπάρχουν υπάρχει δυνατότητα για τέτοια ε, δημοψηφίσματα, αλλά δεν θα έχουν την απαραίτητη νομική βάση ε, ε, και εν πάση περιπτώσει είναι θέμα και διεθνούς δικαίου και ευρωπαϊκού δικαίου. Δεν είναι δυνατόν να πει κανείς ότι ένα δημοψήφισμα της, που γίνεται, που οργανώνεται σε μία χώρα μέλη θα πρέπει να σχετίζεται με, την, με τις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα είναι αρκετά σαφές. Εάν δει κανείς, ας πούμε, το άρθρο 48 ε, σχετικά με την αναθεώρηση των συνθηκών αναφέρει ότι ε, σε σχέση και με τις και σε σεβασμό των, των απαιτήσεων ε, των, των εθνικών συνταγμάτων και των προβλέψεων για δημοψήφισμα. Αλλά όταν αυτό δεν αναφέρεται στο Σύνταγμα και αυτό δεν είναι πολιτικό ζήτημα, είναι συνταγματικό. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει η με τη διαδικασία. Ως νομικό ζήτημα ε, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί αντίθετα από το θέμα των συνθηκών για το άρθρο 48 και επίσης ε, αναφέρονται και οι ε, διατάξεις, ε, γενικές διατάξεις Πασχέλ. Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται και αυτό, δηλαδή νομίζω ότι μπορεί κανείς να ερμηνεύσει βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου και του διεθνούς δικαίου, οφείλει να, να ερμηνεύσει συγγνώμη, το άρθρο 48 με συγκεκριμένο τρόπο και επομένως εάν θέλει ε, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο να, το Ηνωμένο Βασίλειο να ε, εισάγει ζήτημα δημοψηφίσμα, θα να το κάνει σύμφωνα με το άρθρο 48 και βάσει της χρήσης της, της προσωπικής ρήτρας Πασχέλ Υπάρχει επίσης και ένα ισχυρό επιχείρημα το οποίο ε, αναφέρεται ε, από αυτούς που πιστεύουν ότι θα πρέπει να, να καταργηθούν τα δημοψηφίσματα κατά αυτήν την έννοια όσον αφορά ε, το παράδειγμα της Γαλλίας. Είναι εγωιτευτικό το παράδειγμα της Γαλλίας. Ναι, είναι συνταγματικό, συνταγματική απέτηση της ε, Γαλλίας ε, και αυτό έχει ενταχθεί ήδη ε, στις συνθήκες από το 2000 και επομένως είναι σαφές ότι μπορεί η Γαλλία να έχει μια τέτοια ποίηση. Τώρα όσον αφορά τις ε, ε, ε, σχετικά ας πούμε με την παρατήρηση ότι στη Γαλλία μπορεί να ψηφιστεί ας πούμε ένα θέμα που αφορά την νομοθεσία στα πλαίσια μιας πρωτοβουλίας ε, πολιτών ε, και αυτή καταψηφιστεί, τότε ε, μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι αυτό θα είχε καταψηφιστεί και σε μια συνήθη νομοθετική διαδικασία, στο Συμβούλιο δηλαδή. Κατά αυτή την έννοια Ε, θα πρέπει να συζητηθεί μεν, αλλά μπορεί να έχει και μια νομική βάση κατά την έννοια που ανέφερα προηγουμένως. Υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες που δεν είναι ε, επικαιροποιημένες. Ναι, αυτό που είπε και η κυρία Πρόεδρος, στο ερώτημα που έθεσε, ε, είναι γεγονός ότι δεν έγιναν οι μεγάλες αλλαγές οι οποίες θα έπρεπε ε, ε, μπορούν όμως να υπάρξουν τροποποιήσεις όσον αφορά ε, το, την πρωτοβουλία των πολιτών. Ναι, μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω το θέμα στις συνθήκες. Όσον αφορά τώρα δεύτερο δημοψήφισμα, κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι σωστό γιατί όταν κάποιος ε, όταν κάποιος ε, ας πούμε στην Νορβηγία ε, θεωρήσει ότι δεν θέλει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τον υποχρεώνει κανείς όταν η Σουηδία αποφάσισε οι Σουηδοί λένε ότι δεν θέλουν να είναι μέλος της ενιαίας του ενιαίου νομίσματος δεν έγιναν μέλη του ενιαίου νομίσματος είναι πάρα πολύ δύσκολο και έχει ασκηθεί σημαντική αρνητική κριτική σε αυτή την ιδέα των δευτέρων δημοψηφισμάτων Νομίζω πως ε, οι συνάδελφοι κάλυψαν τα περισσότερα θέματα. Θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Ε, είναι λίγο λάθος το όνομα. Δεν είναι μία πρωτοβουλία πολιτών, είναι μία ε, πρωτοβουλία που είναι ανάμεσα στην απόλυτη άμεση δημοκρατία που συλλέγει υπογραφές και στο τέλος έχει ένα αποτέλεσμα και σε ένα ε, αντιπροσωπευτικό σύστημα. Είναι σπάνιο, αλλά δεν είναι ανήκουστο. Για ένα παρόμοιο πολιτικό σύστημα, όχι ακριβώς το ίδιο με τις Ευρωπαϊκές Ένωσης, αλλά με ένα ομοσπονδιακό σύστημα. Υπήρξαν λοιπόν ορισμένες περιπτώσεις που είχαμε πρωτοβουλίες θεματικές, Αργεντινή, Βραζιλία, Αυστρία για παράδειγμα, χώρες με ομοσπονδιακέ δομές, ε, πρωτοβουλίες οι οποίες είχαν ένα συγκεκριμένο θέμα, δεν οδήγησαν όμως σε κάποιο αποτέλεσμα. Είχαν όμως, αν όχι άμεσες επιπτώσεις, έμεσες επιπτώσεις. Είχαμε, όπως είπατε και εσείς, πάνω από 50 τέτοιες πρωτοβουλίες πολιτών και έτσι συγκριτικά είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών έχει το όνομα κατά Δεν είναι ακριβώς πρωτοβουλία πολιτών. Είναι μία ταμπέλα αν θέλετε η οποία βέβαια δεν είναι θετική ή αρνητική. Είναι ακριβώς όπως ε, λέει κάποιος ότι είναι αριστερός ή δεξιός. Έχει οικονομική ιδεολογία ή συγκεκριμένες προτιμήσεις για το ρόλο του κράτους. Τώρα, ο φόβος και ο θυμός που είπατε πολύ σωστά είναι κάτι που πρέπει να συνηθίσουμε. Είναι κάτι που είδαμε στα περισσότερα πρόσφατα δημοψηφίσματα και είναι μάλιστα και ένας στόχος των όσων διεξάγουν το δημοψήφισμα να δημιουργήσουν φόβο το εκλογικό σώμα, έτσι ώστε να διατηρηθεί, να αλλάξει το status quo. Είναι δηλαδή μια προεκλογική στρατηγική, η οποία βέβαια δεν έχει πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως είδαμε, είτε με την περίπτωση του Brexit, είτε με το ελληνικό δημοψήφισμα. Δεν ε, υπολόγιζαν ε, κάποιοι στον θυμό των πολιτών. Μετά, ε, σε σχέση με τη Γαλλία και το δημοψήφισμα, να σας πω ότι οι περισσότερες χώρες που διεξάγουν δημοψηφίσματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση μοιάζουν πάρα πολύ με την ε, περίπτωση της Γαλλίας. Ελάχιστα δημοψηφίσματα ε, προκλήθηκαν και διεξήχθησαν ως άμεσο αποτέλεσμα του συντάγματος μια χώρας ακόμα και αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ρήτρα η οποία θα θέτει σε ισχύ την διεξαγωγή δημοψηφίσματος, έχουν γίνει τα δημοψηφίσματα όπως σας είπα. Επίσης δεν υπάρχουν τόσες πολλές πρωτοβουλίες από κάτω προς τα πάνω όπως έγινε στην περίπτωση της Ολλανδίας από αυτή την ομάδα ευρωσκεπτικιστών. Επίσης, μην ξεχνάμε το ρόλο των μέσων ενημέρωσης, ο οποίος ολοένα και αυξάνεται και ολοένα και αυξάνει την επιρροή του το στάδιο της συλλογή υπογραφών. Πρέπει να δούμε λοιπόν τα μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα τα κοινωνικά ε, μέσα, σε σχέση με αυτές τις ε, πρωτοβουλίες βάσης. Μετά μιλήσατε και για τον Δήμο. Ο Δήμος δεν είναι προϋπόθεση για ένα δημοψήφισμα. Η Ελβετία, για παράδειγμα, δεν έχει Δήμο, δεν έχει τέτοιο σώμα. Έχει κάποιες κοινότητες, τρεις-τέσσερις, οι οποίες είναι μικρές πολλές φορές. Δεν είναι λοιπόν απαραίτητη προϋπόθεση αυτή. Μετά, τι άλλο έχω σημειώσει. Ναι, και ένα ευρύτερο ζήτημα για την άμεση δημοκρατία. Ακούστηκαν κάποια σχόλια πως υπάρχει δυσπιστία απέναντι στα μέσα άσκησης άμεσης δημοκρατίας και για πολλούς εύλογους λόγους. Όμως, εάν βγάλουμε όλες τις λεπτομέρειες και μείνουμε στην ουσία, θα δούμε ότι συνοψίζεται το κύριο επιχείρημά του στο ότι ο απλός κόσμος δεν είναι σε θέση να καταλάβει τόσο πολύπλοκα ζητήματα, δεν θα έπρεπε η άμεση δημοκρατία να είναι τόσο άμεση κτλ. Βέβαια, ε, αν το πούμε αυτό για το δημοψήφισμα, τι θα κάνουμε στην περίπτωση των εκλογών. Βέβαια, νομίζω πως Είδαμε σαφέστατα χθε ότι όταν ο κόσμος ψηφίζει σε ένα δημοψήφισμα δεν ψηφίζει απαραίτητα για το θέμα ε, για το οποίο ερωτάτε, αλλά ψηφίζει πολιτικά, όπως είδαμε με την Ιταλία χθε το βράδυ. Οι περισσότεροι ψήφισαν για την πολιτική του Ρέντσι παρά για το ε, θέμα που ε, είχε το δημοψήφισμα. Βέβαια, οφείλουμε να ρωτήσουμε αυτούς και το εξής. είναι το θέμα του ποιο κόμμα ε, μας εκπροσωπεί καλύτερα σε εκλογές. Όχι, πολλοί ψηφίζουν σε εκλογές ακριβώς ε, επειδή θεωρούν ότι ο ηγέτης είναι χαρισματική φυσιογνωμία και όχι επειδή το πρόγραμμα του κόμματος τους εκφράζει. Η δημοκρατία μας λοιπόν δεν είναι τέλεια, δεν μπορεί να είναι τέλεια, δεν υφίσταται τέλεια, η άμεση, τέλεια άμεση δημοκρατία όπως είπατε. Ακόμα και στην Ελβετία δηλαδή, το η, οποία οποίας η περίπτωση είναι ό,τι πιο κοντινό στην άμεση δημοκρατία, είναι σχεδόν ας πούμε άμεση δημοκρατία, με διαμεσολαβητές στα πολιτικά κόμματα, ακόμα και ε, ένα δημοψήφισμα στην Ελβετία, αν περάσει, υπάρχουν πολλά στάδια μέχρι να φτάσει στην εφαρμογή, όπως για παράδειγμα το, για το δημοψήφισμα με τις ποσοστώσεις ε, μεταναστών. Μετά η, η Ελλάδα ήταν μια άλλη περίπτωση το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου για τον Brexit. Δεδομένης τη αλληλεξάρτηση που ανέφερε ο καθηγητή Ρόουζ, είναι πολύ δύσκολο να εφαρμόσουμε την απόφαση ενός δημοψηφίσματος, ακριβώς ε, παίρνοντας παράδειγμα τα τρία δημοψηφίσματα που προανέφερα. Σα ευχαριστώ. Ναι, να πω κάτι σύντομο καταρχάς. σε ένα δημοψήφισμα, ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιστραφεί το αποτέλεσμα και μάλιστα γύρονται και περισσότερα θέματα μετά από ένα δημοψήφισμα τα οποία είναι σχετικά σε αυτό. Ένα από αυτά τα θέματα στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν και ε, η αποχώρηση. Τώρα η Τερέζα Μέι είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και ε, όσο και αν υπάρχει επιθυμία να προσπαθήσει να βρει μια εναλλακτική λύση, ένα συμβιβασμό, όχι, μέσα σε δύο χρόνια πρέπει να ενεργοποιήσει το άρθρο 50. Φανταστείτε τι θα γίνει. Ε, όμως, η Σκοτία είναι μια εξαιρετική περίπτωση, διότι στην ε, περίπτωση του δημοψηφίσματος είναι η μόνη οντότητα που μπορεί να ανατρέψει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Βέβαια, η συνθήκη είναι μια συνθήκη που υπογράφεται μεταξύ κρατών και όχι μεταξύ ανθρώπων. Και εδώ περνάμε πάλι σε αυτό που λέγαμε πιο πριν, ότι σε μια βασιλεία όλοι είναι υποτελεί σε ένα βασιλιά, ο οποίος δεν εκλέγεται. Υπάρχει κληρονομική διαδοχή και εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα του τι είδους διακυβέρνηση επιθυμούν οι πολίτες. Μετά, αν κοιτάξουμε τα συντάγματα διαφόρων χωρών, θα δούμε πως όλα έχουν προβλέψει δυνατότητα τροποποίησης. Πολλές φορές αυτές οι διατάξεις είναι κρυμμένες, είναι θέμα ερμηνείας, αλλά σκοπός τους είναι να μην υπάρχει οπισθοχώρηση, να κοιτάζουμε προς τα μπροστά. Τα δημοψηφίσματα λοιπόν είναι ένα είδος αντίδρασης. Ένα είδος αντίδρασης για θέματα εθνικά κυρίως, αλλά και όπως έχουμε δει υπερεθνικά. Και είδαμε επίση και τα πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν από αυτέ τι επιλογέ. Εγώ θέλω να σταθώ στο εξή. Από τη μία χρειάζεται να προσπαθήσουμε και μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συσπυρώσουμε δυνάμεις, να ενημερώσουμε, να βεστιτοποιηθούμε. διότι εάν εσείς οι ευρωβουλευτές ε, ευαισθητοποιηθείτε και προσπαθήσετε να ενημερώσετε τους ψηφοφόρους σας, τότε πιστεύω πως θα έχουμε πρόοδο. Μετά υπάρχουν και αντεπιχειρήματα σε ένα δημοψήφισμα. Αντεπιχειρήματα ενός ε, αποτελέσματος το οποίο ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Υπάρχουν προβλήματα αλληλεξάρτησης τα οποία πρέπει να λυθούν, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση το πρόβλημα του νομίσματος, του δανεισμού, της μετανάστευσης, οικονομικών μειονεκτημάτων, μειονεκτήματα ανταγωνισμού μετά από μια αποχώρηση. Θα υπάρχουν προβλήματα, ό,τι και αν γίνει. Και μάλιστα δεδομένων αυτών των περιορισμών που προκύπτουν από τις εθνικές σε δημοκρατίες και από τους πλουραλιστικές υπερεθνικές δημοκρατίες είναι αναγκαίο να δούμε ξανά το γιατί ψηφίζουν οι πολίτες. Αλλά το θέμα είναι επίσης και ποια πολιτική είναι αποτελεσματική. Πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να θυσιάσεις κάτι για να κερδίσεις κάτι άλλο. Στην προκειμένη περίπτωση να θυσιάσεις λίγη εθνική δημοκρατία για να κερδίσεις κάτι μεγαλύτερο. Ε, στη μετανάστευση για παράδειγμα. Αυτό όμως που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην θυσιάσουμε εθνική κυριαρχία, εθνική δημοκρατία χωρίς να κερδίσουμε κάτι που θα ε, ωφελεί περισσότερου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σμοντάλβο. Πολύ σύντομα. Πιστεύω ότι ήδη υπόθηκαν πάρα πολλά. Είναι σαφές ότι υπάρχουν κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά κράτη και η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και βεβαίως το Ηνωμένο Βασίλειο ε, ε, έχει ένα πολύ ειδικό πλαίσιο το οποίο δεν μπορεί να να εφαρμοστεί σε άλλες χώρες ε, και ε, έχω να πω ότι, ε, και το λέω με πολύ μεγάλη αγάπη και εκτίμηση για το Ηνωμένο Βασίλειο, ότι στην ουσία το 2011 αποποιήθηκε κατά κάποιο τρόπο το πραγματικό του κοινοβουλευτικό σύστημα. Επίσης δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν οι κανόνες στο θέμα της, στο θέμα της Σκοτίας ε, ήταν λίγο, αν μου επιτρέπετε, ε, λίγο το πέναλτι το οποίο το χτυπάμε και το ξαναχτυπάμε, και μας αφήνουν μέχρι να βάλουμε τον γκολ. Ε, το ζήτημα είναι ότι όταν χτίζεται ένα σύστημα το πρώτο είναι να καλυφθούν ε, οι βασικές θεμελιώδεις αρχές και τα θεμελιώδη δικαιώματα των μειοψηφιών. Στην περίπτωση βέβαια των δημοψηφισμάτων τα δικαιώματα των, των μειοψηφιών ε, καταπατούνται. Ε, σε σχέση με το δημοψήφισμα της Ιταλίας πιστεύω ότι είναι από τα πιο αποδεκτά. Δηλαδή στην ουσία γίνεται μια προσπάθεια περιορισμού των δημοψηφισμάτων, ε, ε, λαμβάνοντα υπόψη ε, όλα τα, τα στοιχεία πολιτικά και συνταγματικά. Εγώ παρακολούθησα το δημοψήφισμα της Ιταλίας που εν μέρει ακολούθησε το περιφερειακό ισπανικό πρότυπο. Το δημοψήφισμα της Ιταλίας είναι πολιτικό και ε, ε, συνταγματικό και δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε ε, αυτού του είδους το δημοψήφισμα και αφορά το πλαίσιο της Ιταλίας καθορίζοντας λοιπόν κάτι σε επίπεδο μιας χώρας καθορίζεται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης εγώ βέβαια βλέπω ότι θα μπορούσε να οδηγήσει ότι το κίνητρο είναι η αποφυγή αστάθειας πράγμα που είναι κακό και για την ίδια χώρα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το, το ζήτημα είναι ε, να μην προσφύγει κανείς σε ευρωπαϊκό ε, δημοψήφισμα ή σε δημοψήφισμα γενικά έτσι ώστε να λύσει εσωτερικά προβλήματα. Θα πρέπει τα δημοψηφίσματα να παραμείνουν σε εθελούσια βάση και ε, μη δεσμευτικά όπως είναι στη Γαλλία ε, γιατί διαφορετικά θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα στα συνταγματικά δικαστήρια των ε, κρατών μελών. Υπάρχουν διαφορετικές μορφές δημοψηφίσματος. Το δημοψήφισμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ότι η Ευρώπη είναι ένα περίεργο είδος. Μιλάμε για κάτι διαφορετικό και μιλάω για, τα ε, άποψη νομική και συνταγματική. Δεν είναι, κάτι, δεν είναι ένα είδος κοινό στις δημοκρατίες μας. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να ε, υπάρχει μεγαλύτερη διοκτησία και μεγαλύτερη συμμετοχή. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει την δυνατότητα, έχει ξεκινήσει μια σκέψη ε, για ε, ε, ε, συζήτηση, ε, κάποιες, κάποια πρότυπα επίσης συμμετοχής στο νομικό, στη νομική διαδικασία υπάρχουν πολλές εκτός από την προσφυγή σε δημοψήφισμα το οποίο ακριβώς λόγω της δομής του και της απάντησης ναι ή όχι μπορεί να απαγορεύσει κάποιες λύσεις και οπωσδήποτε να καταπατήσει τα δικαιώματα της μειοψηφίας αν θέλουμε μια πραγματική αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ε, ε, μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία νομίζω ότι μπορούμε να ε, λειτουργήσουμε με τον τρόπο τον οποίο έχουμε λειτουργήσει μέχρι τώρα. Ναι, ότι απομακρύνονται οι πολίτες είναι αλήθεια γιατί ε, υπάρχει μια, μια ε, απομάκρυνση λόγω της κρίσης. Μετά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο βλέπουμε ότι για πρώτη φορά δεν γίνονται σεβαστές αυτές οι αρχές της αδελφότητας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και επομένως ε, νομίζω ότι αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουν ενταθεί λόγω της κρίσης θα πρέπει να τα λύσουμε με, μέσω, ε, ε νομικών και συναματικών λύσεων και όχι μέσω δημοψηφισμάτων και πολιτικών λύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Λέει η Πρόεδρος. Ε, ολοκληρώσαμε λοιπόν τη συζήτηση. θα σας παρακαλούσα να μας στείλετε και κάποια, κάποια γραπτά ε, θέματα τα οποία αφορούν την, ε, τις ε, παρουσιάσεις σας, έτσι ώστε να τα βάλουμε και εμείς στα δικά μας στις δικές μας ιστοσελίδες. Σε δύο λεπτά θα ξεκινήσουμε την επόμενη συζήτηση που είναι η παρουσίαση του κυρίου Charles Grant και που αφορά το Brexit. Δύο λεπτάκια διακοπή παρακαλώ.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 Συνάδελφοι, ξεκινάμε. Αν θέλετε, τα πηγαδάκια να μεταφερθούν εκτός της αίθουσας. Κάποιοι θα θυμάστε ότι η πρώτη συζήτηση στην Επιτροπή μας για ε, τις επιπτώσεις του Brexit έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου 2015. Τότε είχε έρθει πάλι ο Charles Grant και τότε μας μιλούσε για ένα πιθανό Brexit που βέβαια φαινόταν ότι απήχε πολύ από την πραγματικότητα. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει δραματικά. Όμως ε, να πω δύο λόγια πριν ε, δώσουμε το λόγο στον Charles για να του δώσω και λίγο μια αίσθηση ε, του κλίματος, της ατμόσφαιρας εδώ. Όλο ένα και περισσότερα εξετάζουμε ένα πιθανό Brexit σαν ένα από μια σειρά ζητημάτων που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώ και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, είμαστε διατεθειμένοι να παρακολουθήσουμε και του σύνεγγυ στη διαδικασία του ώστε στο τέλος ε, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, στο τέλο των διαπραγματεύσεων, και για την επίτευξη της τελικής συμφωνίας ε, να ε, προετοιμάσει μια σύσταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υπερψηφίσει ή να καταψηφίσει η Ολομέλεια. Θα είμαστε λοιπόν αρμόδιοι για την ε, συγκατάθεση ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό συνεχίζουμε τις, και θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις από τώρα μέχρι και το τέλος των διαπραγματεύσεων για να έχουμε μια συνολική επισκόπηση της κατάστασης και να μην μας, ξεφύγουν στοιχεία που είναι σημαντικά για την τελική θέση και στάση του Κοινοβουλίου. Όλο ένα και περισσότερο όμως αναγνωρίζουμε τους κινδύνους που ελοχεύουν στην όλη διαδικασία. Ανησυχούμε ότι μπορεί να υπάρχει και η πιθανότητα η διαδικασία ε, να παρουσιάσει καθυστερήσεις, να μην είναι τόσο ταχεία όσο θα περίμενε κανείς, γιατί εν τω μεταξύ για τις δύο ε, όχθες ε, της μάχης ο καθένας ε, αναπτύσσει τα δικά του μάντρα και μότο. υπάρχει λοιπόν μια αίσθηση από την Βρετανική πλευρά ότι η Ευρώπη θα τους δώσει αυτό που θέλουν. Από την άλλη στην Ευρώπη λέμε ότι κανείς εκτός Ευρώπης δεν μπορεί να έχει καλύτερες, καλύτερους όρους και προϋποθέσεις από ό,τι τα κράτη-μέλη. Επομένω, ε, το χάσμα μεγαλώνει. Δεν γεφυρώνεται και πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να λάβουμε υπόψη και αυτή την πρόκληση ως πολιτική. Ε, μακάρι να με διαψεύσετε για αυτούς τους κινδύνους και για τα χάσματα. Σας δίνω το λόγο, έχετε όσο χρόνο θέλετε, αλλά κατά νου είχαμε μια παρέμβαση 15 λεπτών και μετά να γίνει μια συζήτηση μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που επιστρέφω σε αυτή την Επιτροπή. Θα ήθελα ε, να περιγράψω πώς εγώ ε, βιώνω το Brexit ε, από βρετανικής πλευράς. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο δυνατόν πιο αντικειμενικός και μετά θα πω και δύο λόγια στο τέλος για την Σκοτία, την Ιρλανδία και τα νομικά, τη νομική υπόθεση ενώπιον του του Δικαστηρίου που ξεκίνησε σήμερα. Αρχικά να πω γιατί θα είναι αρκετά σκληρό το Brexit. Δηλαδή εννοώ ότι η τελική συμφωνία θα οδηγήσει σε σημαντική ε, μείωση των εμπορικών και οικονομικών ε, ε, σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας από τους λόγους είναι ότι το πολιτικό κατεστημένο ζει ακόμα σε μια μικρή φούσκα. Επειδή η οικονομία δεν έχει πληγεί ουσιαστικά, έχουν πιστέψει κάποια από τα επιχειρήματά τους ότι μπορούν να έχουν και την πίτα και το σκυλοχορτάτο δηλαδή χωρίς να πληγεί η οικονομία τους, ε, να ε, κόψουν ε, τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πολιτικό υπόβαθρο. Επίσης, πρέπει κατά τη γνώμη μου να επισημάνουμε ότι αυτό είναι μια λανθασμένη άποψη. Η Βρετανική θέση είναι μάλλον ε, αδύναμη. Ξέρετε για το άρθρο 50 ότι έχουμε 50, ε, συγγνώμη, δύο χρόνια για να εκκινήσουμε τη δικασία του άρθρου 50 και αν υπάρξει μια διευθέτηση μετάβασης, αν υπάρξει τέτοια λοιπόν. Ιδάλλως, ε, αν δεν καταφέρουμε να κλείσουμε μια τέτοια συμφωνία δύο, στα δύο έτη, μπαίνουμε στου κανόνε του ΠΟΕ. Πρέπει να υπάρχει όμω ε, καλή βούληση από του εταίρου. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει καλή συμφωνία. Και δυστυχώ οι επαφέ ε, του τελευταίου μήνε δεν ήταν πολύ θετικέ. Για παράδειγμα, ο Μπόρι Τζόνσον ανέφερε ότι η ιδέα τη ελεύθερη ε, κυκλοφορία ω θεμελιώδου αρχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια σχέτη βούρδα. Αυτό είπε. Και αυτή δεν είναι μοναδική τέτοια περίπτωση που έχω κατά νου. Άλλο γεγονό, υπάρχει η μεγάλη αναστάτωση ε, στο κόμμα των εργατικών. Το κόμμα δεν έχει ισχυρή ηγεσία, υπάρχει σημαντικό ε, διχασμό για το τι θα πρέπει να γίνει. Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών, που είναι το πλέον ισχυρό Υπουργείο στο Βρετανικό σύστημα, είναι πολύ πιο αδύναμο από ό,τι συνήθω ε, από την εποχή του Μπλέρ ή του Κάμερον, α πούμε παρότι ο Χάμοντ είναι αρκετά ε, λογικός άνθρωπος και πολιτικός, ε, νομίζω ότι μεγάλη εξουσία, πολλή εξουσία συγκεντρώνεται ε, στο Πρωθυπουργικό Γραφείο όπου δεν υπάρχει μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη για το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω αυτό να επιληθεί αρκετά σύντομα. Κλείνοντα, τελευταίο λόγο για τον οποίο θεωρώ ότι δεν θα πάνε καλά τα πράγματα για τον Brexit. Ο επιχειρηματικός κόσμος που βέβαια είναι υπέρ ενός ήπιου Brexit, δεν έχει ε, βρει ακριβώς τον τρόπο να ασκήσει πιέσεις. Ε, μιλούν ε, με τα διάφορα υπουργεία, όμως η κυβέρνηση των συντηρητικών δεν ενδιαφέρεται απαραίτητα και τόσο πολύ για τις απόψεις τους παρότι συνήθως οι κυβερνήσει των συντηρητικών είναι υπέρ των επιχειρηματιών συνήθως. Τέλος, ε, ε, ο κίτρινος τύπος είναι πολύ ισχυρός και αυτό το έχουν επισημάνει και βεβαιώσει πολλοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Η κυβέρνηση λοιπόν φοβάται ότι ο κίτρινος τύπος ε, θα ε, τους κατηγορήσει ότι έχουν ε, προδώσει τη βούληση του λαού αν πάνε και επιλέξουν ένα ήπιο Brexit γιατί θεωρείται ότι έχουν ψηφίσει οι Βρετανοί για ένα ε, σκληρό Brexit, ενώ στην ουσία ψήφισαν για ένα Brexit. Πρέπει λοιπόν ε, να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με τις, ε, τους οικονομικούς δεσμούς της Μεγάλης Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα είπα όλα αυτά. Βέβαια υπάρχουν και λιγότερα απεσιόδοξε απόψεις. Εδώ στις Βρυξέλλες πολλοί θεωρούν ότι θα είναι πολύ δύσκολο το Brexit. Άλλοι θεωρούν ότι θα, δεν θα υπάρξει καν μεταβατική τέτοια περίοδο. Εγώ γιατί είμαι λιγότερο απεσιόδοξο. Γιατί θεωρώ ότι η οικονομία ε, θα πληγεί, μπορεί να διαψευστώ, όμω θεωρώ ότι θα πληγεί σύντομα. Ξέρω ότι πολλέ επιχειρήσει ε, αναβάλουν ή ακυρώνουν επενδύσει. Πολλέ ε, τέτοιε κινήσει έχουν γίνει ε, μακριά από τα φώτα τη δημοσιότητα. Υπάρχει μια πλειοψηφία ε, υπέρ της ε, του, του ήπιου Brexit ε, στην ε, Βουλή των Κοινοτήτων. Και θεωρώ ότι και η Πρωθυπουργό ε, ίσως ξεκινά από διαφορετική οπτική γωνία. Διαβάζει πάρα πολύ εντατικά για το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι μαθαίνει πολλά πράγματα. Και κάποια στιγμή θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρει αποστάσεις από την δεξιά πτέρυγα των συντηρητικών και να πει αυτή τη συμφωνία θέλω και θα είναι μια συμφωνία που θα καταπλήξει όσους ήθελαν ένα πιο σκληρό Brexit. Αυτό πιστεύω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος. Τώρα, τι αναμένουμε. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι η μεταβατική συμφωνία για τους εμπορευόμενους στη Βρετανία. Αυτό προφανώς γιατί θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον το 2019, ε, η μελλοντική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών θα τεθεί σε ισχύ ίσως μετά από μια πενταετία, όταν θα έχει εγκριθεί ε, από τα κοινοβούλια κτλ. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια μεταβατική συμφωνία. Το πρόβλημα για την κυρία Μέη, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ και έχετε και τη δικιά σα πηγέ εδώ, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πολύ σκληρή σε ό,τι αφορά τι ε, ε, προβλέψει, τι διατάξει θα δεχτείτε ε, την ελεύθερη κυκλοφορία, τη αποφάση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλιώ δεν θα πάρετε μεταβατική συμφωνία. Όμω θα πρέπει ίσω να είναι οι Βρετανοί πιο ευέλικτοι από ό,τι θα ήθελαν. Δεν είμαι σίγουρο ότι θα είναι. Θα υπάρξει νομίζω μεταβατική συμφωνία. Νομίζω ότι οι Βρετανοί θα θέλουν μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ε, στυλ Καναδά, Καναδά Plus. Να έχουν δηλαδή μεγαλύτερη πρόσβαση ε, στην ευρωπαϊκή αγορά υπηρεσιών σε σχέση με τον Καναδά. Όμω ε, δεν θεωρώ ε, να ζητά κανείς διαβατήριο για να πάει στο Λονδίνο. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς ε, θα επιτρέψουν σε ε, τράπεζες στο ΣΥΤΙ να δραστηριοποιούνται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς κανένα περιορισμό. Δεν νομίζω ότι θα είναι διατεθειμένη η Αγγλία να δεχθεί την ελεύθερη κυκλοφορία και τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Γι' αυτό δεν θα είναι στην εσωτερική αγορά ούτε τελωνιακή ένωση. Κατά πάσα θεωρώ δεν θα γίνει ούτε αυτό. Νομίζω ότι η Βρετανία θα καταβάλει σφορά στον ευρωπαϊκό προπολογισμό και ο Ντέβιν Ντέιβις το ανέφερε πριν από μερικές ημέρες στη Βουλή και σε ό,τι αφορά τους περιορισμούς ως προς την ελεύθερη κυκλοφορία που σίγουρα θα εφαρμόσει η Βρετανία νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επιβάλλουν οι περιορισμού περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία για του Ευρωπαίου πολίτε σε σχέση με ε, πολίτες τρίτων χωρών. Ξέρω ότι κάποιοι υπουργοί ε, είναι υπέρ τη διαφοροποίηση μεταξύ Ευρωπαίων και άλλων πολιτών. Αλλά αυτό δεν είναι σίγουρο θα περάσει. Από την άλλη, θεωρώ ότι ο περιορισμό στην ελεύθερη κυκλοφορία θα ε, είναι μια σοβαρή προσπάθεια περιορισμού των του αριθμού ε, των Ευρωπαίων που έρχονται να εργαστούν στον Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό με οδηγεί στο επόμενο. Αντίκτυπο στην οικονομία. Σίγουρα θα το διαρευνάτε και ξεχωριστά. Όμω θεωρώ ότι ένα από το κόστος είναι, ε, τα κόστη είναι ότι οι εργοδότες δεν θα βρίσκουν τόσο εύκολα εργαζόμενους Δεν υπάρχει ανεργία. Είναι 4,7-4,8% στην Βρετανία ενέργεια αυτή τη στιγμή. Αν υπάρξει σημαντικό περιορισμό τη ευρωπαϊκή μετανάστευση, αυτό θα δημιουργήσει πολύ σημαντικό πρόβλημα στην, ε, στον κλάδο των ξενοδοχείων, στη γεωργία, στον επιστημισμό, στι επενδυτικέ τράπεζε, στα think tanks, στο NHS και ούτω καθεξής. Και αυτό είναι ένα μακροπρόθεσμο κόστος προς την ε, βρετανική οικονομία. Ένα άλλο, ακόμα μεγαλύτερο, θα είναι η ε, απώλεια των ε, άμεσων ξένων επενδύσεων. Ξέρω πολλές επιχειρήσεις που έχουν αποφασίσει να μην χτίσουν εργοστάσια και μονάδες ε, στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν θέλουν να το δημοσιοποιήσουν γιατί θα θεωρηθεί μη πατριωτική κίνηση. Αλλά μακροπρόθεσμα ε, η έλλειψη άμεσων ξένων επενδύσεων θα είναι πρόβλημα. Το City θα παραμείνει μεγάλο σημαντικό οικονομικό κέντρο και μετά τον Brexit, όμως σημαντικό τμήμα μερίδιο της αγοράς αυτής θα πάει στη ΣΥΠΑ, στην Ασία, κάποιο θα εξαφανιστεί. Σημαντικό όμως, 10% θεωρώ, θα χαθεί ή θα φύγει μάλλον. Ένα, μια σημαντική επίπτωση θα είναι έλλειψη ε, από όλοι μάλλον φόρων για το Υπουργείο Οικονομικών. Περίπου 60 δις ε, λίρες συμβάλλει το ΣΥΤΙ. Ε, τμήμα του θα χαθεί λοιπόν από αυτή την άποψη. Τέλος, ασφάλεια. Εδώ έχει πιο ισχυρή θέση η Μεγάλη Βρετανία θα υπάρξει ε, σκληρή στάση λοιπόν από τους Ευρωπαίους για το οικονομικό σκέλος, γιατί δεν θέλουν να δουν τη Μεγάλη Βρετανία να ανθίζει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αν υπάρξει αυτή η εικόνα, κάποιοι ευρωσκεπτικιστές θα πούνε ορίστε, μια χαρά τα πήγαν και οι Βρετανοί, ας κάνουμε και εμείς το ίδιο. Επομένω, στα οικονομικά θα είναι πολύ σκληρή. Στα θέματα ασφάλεια θα είναι όμω πιο ήπιοι, γιατί έχουν πολλά να προσφέρουν οι Βρετανοί. Πολλά που χρειάζονται οι Ευρωπαίοι πολύ καλούς διπλωμάτες, ε, κατασκόπους, ε, στρατιωτικούς, ε, τεχνογνωσία για την αντιτρομοκρατία, αστυνομία. Επομένω, αν είναι τυχεροί Βρετανοί, θα μπορούν να καταλήξουν συμφωνία σε αυτού του τομεί που δεν θα του δώσουν θέση στο τραπέζι και δικαίωμα ψήφου, αλλά θα είναι αρκετά κοντά. Το ελπίζω και σίγουρα θα το επιδιώξουν οι Βρετανοί. Κλείνοντα, για τη Σκοτία. περίμενα και πριν από το δημοψήφισμα ε, ένα αρνητικό αποτέλεσμα να οδηγήσει σε αύξηση των απαιτήσεων για ε, δημοψήφισμα στη Σκωτία. Δεν συνέβη αρκετά. Και αυτό γιατί οι Σκοτσέζοι ανησυχούν για την οικονομία του που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη Βρετανική. Αν βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν η Μεγάλη Βρετανία και βγουν οι Σκοτσέζοι από τη Μεγάλη Βρετανία, ε, παρότι θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υπάρχουν ζητήματα συνοριακών ελέγχων μεταξύ Σκοτίας και Αγγλία και θα υπάρχει και πρόβλημα με την ολοκληρωμένη αλυσίδα ε, εφοδιασμού μεταξύ Σκοτία και Αγγλία. Στα σύνορα δηλαδή. Και επειδή είναι τόσο χαμηλέ οι τιμέ του πετρελαίου, οι Σκοτσέζοι μάλλον χρειάζονται τι ενισχύσει ε, των Άγγλων φορολογουμένων που ενισχύουν αυτή τη στιγμή ε, την ε, σκοτσέζικη οικονομία. Βέβαια, αν αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου, θα χαθεί μάλλον και αυτό ο παράγοντα. Η κυρία Στέρτζον λοιπόν βρίσκονται σε δύσκολη θέση γιατί πολλοί στο κόμμα τη θέλουν και άλλο δημοψήφισμα θεωρούν ότι ίσω μπορούν να το κερδίσουν αυτή τη φορά, γιατί ήταν αρκετά κοντά την, την άλλη φορά. Όμω εκείνη είναι αρκετά επιφυλακτική, συνετή γυναίκα, δεν θέλει να βιαστεί, γιατί αν βιαστεί και τελικά δεν πάει καλά, τότε θα έχει προσωπικά πρόβλημα και το κόμμα τη. Επομένω, θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει ε, δημοψήφισμα στη Σκωτία βράχη ή μέσο πρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα όμω μπορεί να υπάρξει. Για την Ιρλανδία τώρα. Είναι πιο μεγάλο ζήτημα για, την, ε, για το Brexit. Είναι μεγαλύτερο πρόβλημα για του Άγγλου δηλαδή δεν θεωρώ ότι ε, θα, υπάρξει, ε, ο ε, έλεγχος διαβατηρίων στα σύνορα. Βόρειας και Νότιας Ιρλανδίας, γιατί δεν θεωρώ ότι ε, θα ε, εισαχθεί ε, τέτοιος κανόνας για τους επισκέπτες σύντομης διαμονής. Όμως υπάρχει ανάγκη τελωνιακών ελέγχων. Αν φύγει λοιπόν η Βρετανία από την Τελωνιακή Ένωση, που είναι πιθανό αλλά όχι βέβαιο, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα αποφύγουμε κάποιους ελέγχους στα σύνορα μεταξύ, εκεί στα σύνορα για να ελέγξουμε τα έγγραφα, τα διαδικαστικά κτλ. Βέβαια υπάρχουν παραλληλισμοί όπως είναι στα σύνορα Σουηδίας, Νορβηγίας. Μπορεί να υπάρχουν ελάχιστα επίπεδα ελέγχων αν υπάρχει αμοιβή εμπιστοσύνη και έτσι να μην υπάρξει τεράστια γραφειοκρατία, όμως θα υπάρξει κάποια παρουσία στα σύνορα. Οι Ιρλανδοί τα γνωρίζουν καλύτερα από μένα, αλλά την τελευταία φορά στο Δουβλίνο μου είπαν ότι του προβληματίζει οποιαδήποτε φυσική παρουσία στα σύνορα, γιατί θα ήταν ε, ε, μια πρόκληση προς τους τρομοκράτες να ανατινάξουν ή να κάψουν κτλ. Είναι λοιπόν σοβαρό πρόβλημα. Και η ίδια η ειρηνευτική διαδικασία, θα σας πούν οι Ιρλανδοί, ότι εξαρτάται από την ευρωπαϊκή, ε, τη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και για τις δύο χώρες. Η Ιρλανδική οικονομία επίσης είναι άμεσα συνδεδεμένη με την Αγγλική, ε, εξαγωγές προς την Αγγλία, προς το Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικά ανεπίλητα ζητήματα. Δύο τελευταίε παρατηρήσει. Δικαστική υπόθεση που ξεκίνησε σήμερα. Λιγότερο ενδιαφέρουσα από ό,τι φαίνεται. Οι περισσότεροι νομικοί θεωρούν ότι το ανώτο δικαστήριο θα ε, πάει ενάντια της κυβέρνησης και να τους πει ότι ε, ενεργοποιείται το άρθρο 50 παρανόμως. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει όμως το Brexit. Έχω μιλήσει και με στηρητικούς ευρωβουλευτές, συγγνώμη, βουλευτές. Οι περισσότεροι είναι κατά του Brexit, θα υπερψηφίσουν όμως την νομοθεσία στο Κοινοβούλιο, γιατί δεν θέλουν να φανεί ότι ε, κινούνται αντίθετα στη βούληση του Βρετανικού λαού θα πούνε θα το υπερψηφίσουμε το νομοσχέδιο, αλλά παρακαλούμε να εκδώσετε μια πράσινη βίβλο που να αναφέρει του στόχου σα. Δεν θα πούνε όχι, εμεί ασκούμε βέτο, δεν ψηφίζουμε το νομοσχέδιο εφόσον εσεί δεν έχετε αναφέρει του στόχου. Πολλοί λοιπόν δεν θα κρατήσουν τόσο σκληρή στάση. Κάποιοι θα καταψηφίσουν το άρθρο 50, Ken Clark και μικρή ομάδα ε, των συντηρητικών θα καταψηφίσει. Ίσως οι φιλελεύθεροι, ε, οι Σκοτσέζοι κτλ. Όμως αυτή είναι 70-80 δεν είναι παραπάνω. Δεν θα σταματήσουν λοιπόν το Brexit, ούτε η Βουλή των Λόρδων θα μπλοκάρει τη διαδικασία. Μίλησα με ορισμένους και δεν θέλουν ε, να φανεί ότι πηγαίνουν αντίθετα με την Βούλη του Βρετανικού Λαού. Δεν θα σταματήσουν λοιπόν, δεν θα μπλοκάρουν τη διαδικασία. Τέλος, ε, υπήρξε στο Ρίτσμοντ ε, ε, εκλεγική διαδικασία όπου η φιλελεύθερη υποψήφια κέρδισε εναντί του συντηρητικού Goldsmith. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει τον Brexit και πάλι, απλώς η συντηρητική θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική. Μέχρι τώρα η κυβέρνηση της κυρίας Μέη είναι ιδιαίτερα επικεντρωμένη στο 52%. Κατά τη γνώμη μου βλέπει και θεωρεί ότι έχει εκλογική εντολή από το δημοψήφισμα να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκληρό Brexit Ε, και να περασπιστεί κυρίως εκείνους που δεν έχουν αποφεληθεί της παγκοσμιοποίησης και που θεωρούν ότι το Λονδίνο ε, τρέχει αυτό το σύστημα και ηγείται χωρίς να του σκέφτεται. Εκλογικά μπορεί αυτό να είναι σοφό, όμως υπάρχουν και ψηφοφόροι ε, συντηρητικών που είναι φιλελεύθεροι και κάτοικοι του Λονδίνου που ψήφισαν για το Brexit. Επομένως είναι πιο σύνθετα τα πράγματα. Ίσως να υπάρχουν 10-15 ε, τέτοιες ε, εκλογικές θέσεις που να ιτηθούν στη Δυτική για ανάλογους ε, λόγους. Πρέπει λοιπόν να σκέφτεται και παραπάνω η κυρία Μέη, όχι μόνο το 52%. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κοινοβούλιο θα μπλοκάρει το Brexit, δεν μπορώ να φανταστώ κάποια νομική, διαδικαστική, κοινοβουλευτική διαδικασία που θα αποτρέψει το Brexit. Κατά τη γνώμη μου, ο μοναδικό τρόπο να επανανταχθεί το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να βγει για μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά να νιώσει αυτή την απομόνωσή τη και να ξαναμπεί. Αλλά αυτό θα πάρει πολύ καιρό. Ευχαριστώ. Uh, thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργη Όπλιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τσάρλς, ε, καλώς ήρθες και χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Έχω μία ερώτηση και θέλω την άποψή σου. Θα γνωρίζεις, φαντάζομαι, το επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι συντηρητικοί ευρωσκεπτικιστές ότι τώρα θα απελευθερωθεί η Βρετανία από τα δεσμά της, θα γίνει η Σιγκαπούρη της Ευρώπης, θα συναλλάσσεται με όλο τον κόσμο κτλ. Είναι εφικτό αυτό, μπορεί να γίνει. Μα ανέφερε ποσοστά και τα λοιπά, αλλά οι εμπορικές και τα ποσοστά των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω αν δούμε τα πράγματα σε έναν κύκλο 7-10 ετών είναι εφικτό να συμβεί κάτι τέτοιο. Υπάρχουν οι δομέ που να διασφαλίζουν ότι ό,τι και να γίνει η αλυσίδα εφοδιασμού θα συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αυτή η μεταβατική συμφωνία θα είναι τόσο σημαντική όσο προβλέπετε. Έχω τι αμφιβολίες μου βέβαια για το αν η Βρετανία θα γίνει η Σιγκαπούρη της Ευρώπης, αλλά εσύ τι άποψη έχεις. Η απάντηση είναι και οικονομική και πολιτική. Η οικονομική απάντηση είναι ως εξής. Αν δούμε το εμπόριο και τις λεπτομέρειες του υπάρχει το μοντέλο βαρύτητας, έτσι αποκαλείται αυτό. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι εκεί που βρίσκεσαι γεωγραφικά ε, είναι πολύ σημαντικό για το τι εμπόριο θα κάνεις και πόσο. Η γεωγραφική σου θέση δηλαδή επηρεάζει το εμπόριο. Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι αναπόφευκτο το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών συναλλαγών να γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μία αποχώρηση θα οδηγήσει σε μείωση του εμπορίου. Αυτή τη στιγμή τώρα οι εμπορικέ συναλλαγέ με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 50% θα μειωθεί αυτό. Όχι όμω δραματικά. Ακριβώ γιατί το κόστο μεταφορά των αγαθών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν και νομικές ομοιότητε, υπάρχουν ε, πολιτισμικέ ομοιότητε κτλ. Σε γενικέ γραμμέ, λοιπόν μπορώ να πω ότι το εμπόριο με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση θα ε, παραμείνει λίγο πολύ ανεπηρέαστο. Η Ιρλανδία επίσης να πούμε ότι είναι μια, σχέση, μια χώρα η οποία έχει πολύ καλές εμπορικές σχέσεις με το Ηνωμένο Τώρα για το αν θα γίνει η Σιγκαπούρη της Ευρώπης δεν γνωρίζω. Υπάρχουν ορισμένοι που υποστηρίζουν μια πιο θατσερική προσέγγιση, δηλαδή μείωση της γραφειοκρατίας ε, δραστικά μείωση της φορολογίας που αυτό με τη σειρά του θα επιφέρει μια άνθηση της οικονομίας. Όμως δεν έχουν πλειοψηφία γι' αυτό στο Κοινοβούλιο, ούτε καν πλειοψηφία μέσα στους ίδιους τους συντηρητικούς για να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω λοιπόν να περάσει πέραν ε, της απλής ε, πρότασης της ιδεολογίας και πιστεύω μάλιστα πως ε, η Τερέζα Μέη είναι πολύ λιγότερο ευέλικτη, πολύ λιγότερο φιλελεύθερη από ότι ο Κάμερον και ο Όσμπορν. Είναι μάλιστα ε, περιπτώσεις που θεωρώ πως έχει αρκετά αριστερές απόψεις για την οικονομία. Μετά, ε, πρέπει να υπολογίσουμε και την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλο αυτό. Υπήρχαν, όπως γνωρίζετε, ορισμένες διαρροές στους Sunday Times ότι εάν δηλα... απειλούσε η Βρετανία ότι αν δεν δοθούν πλεονεκτήματα θα αυξήσει, θα μειώσει μάλλον την εταιρική φορολογία στο 10% για να προσελκύσει επενδύσεις. Αυτό όμως αποτελεί ε, οικονομικό ντάμπινγκ, κοινωνικό ντάμπινγκ και σίγουρα είναι κάτι που δεν θα παραβλέψει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση στη σύναψη της ε, επόμενης συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά τον Brexit. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπρέσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να πω δύο λόγια όσον αφορά το θέμα της ψήφου του Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι Κανείς από εμά και κανείς από τους Βρετανούς δεν περιμένει να αλλάξει το κοινοβούλιο τη λαϊκή ψήφο. Το ζήτημα το οποίο μου φαίνεται λογικό σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι το Κοινοβούλιο να ε, δώσει διαπραγματευτική εντολή στην κυβέρνηση. Νομίζω άλλωστε ότι αυτή είναι η έννοια της ε, συζήτησης που έχει ξεκινήσει και εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι θα ήταν το πιο λογικό και αυτό θα επέτρεπε, μια και θα υπήρχε η ε, διαπραγματευτική εντολή του Κοινοβουλίου, θα ε, επέτρεπε, λέω, να δει κανεί επί βάσεως θα μπορούσε να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Δεύτερο, ε, τα καλά διαζύγια είναι τα σύντομα διαζύγια, τα γρήγορα διαζύγια. Ε, ε, νομίζω λοιπόν ότι και για το δικό μας συμφέρον, ενδεχομένως και της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά τώρα αναφέρομαι στο δικό μας, το δικό μας συμφέρον λοιπόν είναι να μην υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση μέχρι την έξοδο. Από την άλλη πλευρά πιστεύω ότι και η Μεγάλη Βρετανία ε, θα πρέπει γρήγορα να δει ποια είναι η θέση της απέναντι στη συνθήκη ε, και βεβαίως ε, αν θέλει να επιβάλλει και αυτό το δασμό του 10% θα, θα επιβιώσουμε και με αυτό τι να κάνουμε. Νομίζω ότι καλό θα ήταν εμείς να επικεντρώσουμε την εργασία μας τους επόμενους μήνες στην ανάλυση, την αξιολόγηση και περαιτέρω διευκρίνηση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυρίως στη δική μας Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων θα πρέπει να ε, εργαστούμε έτσι ώστε να βρούμε κάποιο είδος ε, εντολής που θα δώσουμε στους διαπραγματευτές μας. Ίσως δεν θα έχουμε την δυνατότητα και την άδεια να δώσουμε ε, μια πραγματική εντολή, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, ε, ε, εκφράσουμε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να απαντήσουμε σε ορισμένα ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί. Η Ιρλανδία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επανειλημμένα μας έχουν υποβάλει οι συνάδελφοι περιπλοκές που μπορεί να προκύψουν. Θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Επίσης, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δούμε τι θέλουμε εμείς πριν ξεκινήσουμε τη διαπραγματευτική διαδικασία. Και χρόνο, πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπούμε ενδεχομένως και σε ε, κάποια ευαίσθητα ζητήματα τα οποία ακόμα υπάρχουν στο τραπέζι όπως ας πούμε το Γιβραλτάρ. Ε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται λοιπόν με την Ιρλανδία αλλά και κάποια τμήματα του Ηνωμένου ε, Βασιλείου άλλα τα οποία καταψήφισαν το Brexit. Εγώ λοιπόν πραγματικά ε, θα ε, παρακαλούσα να επικεντρώσουμε τη δουλειά μας σε αυτά που είπα. Γιατί όλο λέμε τι θέλουν οι Άγγλοι, τι σκέφτονται οι Άγγλοι. Ωραία, να μας τα πούνε και πιστεύω ότι σύντομα θα μας τα πούνε. Εγώ λέω ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας αντιθέτως στις δικές μας επιθυμίες, στον τρόπο με τον οποίο εμείς θέλουμε να τοποθετηθούμε ε, στην ε, διάρκεια των διαπραγματεύσεων και εξ αρχής να έχουμε μια συγκεκριμένη θέση που θα εκπροσωπεί τα συμφέροντά μας, γιατί νομίζω ότι αυτό μέχρι τώρα το παραμελήσαμε. Ε, μπορεί να υπάρχουν ας πούμε, επιστημονικά συμφέροντα, πολιτιστικά απέναντι στις αγγλικές και πολιτικά απέναντι στις θέσεις των Βρετανών. Αλλά κυρίως εγώ θέλω να δω ποιες θα είναι οι δικές μας θέσεις και ποια θα είναι τα δικά μας συγκεκριμένα συμφέροντα σε αυτή την περίπτωση. Ε, μάλλον να έχουμε και μερικές ερωτήσεις ακόμα και μετά η απάντηση. Richard Κόρμπιν. Ευχαριστώ πολύ, Τσάρλς. Ήσουν πολύ ενδιαφέρον, όπως πάντα. Νομίζω πως μια καθυστέρηση κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το άρθρο 50 δεν θα γίνει ακριβώς μόνο λόγω της ε, δικαστικής προσφυγής, αλλά επειδή πρέπει να γίνει απογραφή όλων των θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπίσουν ε, σε κάθε διαζύγιο, έτσι πρέπει να γίνει. Πρέπει να εξεταστούν όλες οι πτυχές, να λυθούν όλα τα θέματα. Και αυτό το διαζύγιο θα είναι συναρπαστικό. Είναι κάτι που θα δυσκολέψει πάρα πολύ την κυβέρνηση, ακριβώς γιατί είναι διχασμένη για πολλά θέματα. Ανέφερα, αναφέρατε μερικά από αυτά. Θα είμαστε μέσα στην ε, νέα αγορά έξω. Τι θα κάνουμε με τις διάφορες ευρωπαϊκές υπηρεσίες οι οποίες ε, εδράζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα χημικά, για την πολιτική αεροπορία, για παράδειγμα. Είναι πολύ σημαντικές επιπτώσεις ε, του Brexit για τη Βρετανία. Και φυσικά δεν είναι θέμα του ότι αποφασίζεις τι, τι θα κάνεις. Ε, χρειάζεται να γίνει πρώτα μία διαπραγμάτευση. Όμως, όταν κάποια στιγμή η ε, κυβέρνηση ξεπεράσει αυτούς τους ε, σκόπελους με την Τελωνιακή Ένωση και τα λοιπά, για παράδειγμα, ε, θα πρέπει να γίνει κάτι σχετικά με αυτό το διχασμό που υπάρχει στους συντηρητικού. Και τότε αρκετοί από όσους ψήφισαν να αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πούν για μισό λεπτό. Αυτά δεν είναι αυτά που ψήφισα εγώ. Εδώ πέρα πάνε για σκληρό Brexit. Εάν λοιπόν υπάρχει μια αλλαγή στην κοινή γνώμη και νομίζω πως ε, είναι ενδεικτικό το ότι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν δείχνουν κάποια τέτοια αλλαγή περί κατά της μίας ή της άλλης άποψης. Δείχνουν αντίθετα δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει το ίδιο χάσμα με πριν. Δεν έχουν αλλάξει οι απόψεις. Προτού μάλιστα αποκτήσουμε μία πλήρη εικόνα του τι σημαίνει η αποχώρηση. Όμως ε, θεωρείς ότι θα αλλάξει ενδεχομένως η άποψη των βουλευτών. Μας είπες και πιο πριν ότι δεν νομίζεις πως ε, ούτε η Βουλή των Κοινοτήτων ε, ούτε η Βουλή των Λόρδων θα ψηφίσει κατά της αποχώρησης. Θα είναι η τελευταία ευκαιρία βέβαια για εκείνους να θέσουν σε ισχύ μια επανεξέταση της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ενδεχομένως θα μπορούσε να τροποποιηθεί το άρθρο 50 έτσι ώστε να δημιουργηθούν ορισμένες προϋποθέσεις για τις ρεπαγματεύσεις, για παράδειγμα να παραμείνει η χώρα εντός της ενίας αγοράς. Είπε επίσης ότι ε, είναι σκοτεινά, είναι σκοτεινό το μέλλον, υπάρχουν μαύρα σύννεφα στον ορίζοντα. Βλέπουμε όμως ότι οι επιπτώσεις είναι ήδη πάρα πολύ σοβαρές. Η Βρετανία έχασε το τριπλό α στις αγορές δανεισμού και τώρα θα χρειαστεί να δανειστεί ακόμα περισσότερα χρήματα και το κόστος αυτού του δανεισμού θα είναι τεράστιο και πολλά άλλα που μας είπε. Εάν συνεχιστεί αυτό, αν, ε, αυξηθούν οι επιπτώσει, θα υπάρξει κάποια αλλαγή της ε, γνώμης ε, των βουλευτών που, που είναι κατά και εάν ναι, τι νομίζεις ότι μπορούν να κάνουν οι βουλευτές γι' αυτό. Ε, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να κάνω κάποια σχόλια. Μιλάμε για το ε, χρονοδιάγραμμα και το χρονικό πλαίσιο. Για το άρθρο 50 μιλάμε γενικά για τρία χρόνια και όλοι συζητούν και το ε, θέμα ότι κανείς δεν θα θέλει να το παρατείνει μετά τα δύο χρόνια. Αλλά εάν δει κανείς πιο προσεκτικά το τι μπορεί να συμβεί και τι πρέπει να συμβεί ε, μέσα σε δύο χρόνια, ε, αποφάσεις Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, στην ουσία ε, θα πρέπει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ε, ε, πριν από το 2018 και άρα πολύ λίγος χρόνος μένει για τις διαπραγματεύσεις. Δεύτερον, αναφερθήκατε και συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι υπάρχει έτσι, είναι μεγάλη πρόκληση αυτή η ενδιάμεση συμφωνία γιατί αυτή θα είναι πάρα πολύ ε, δύσκολη αλλά και πολύ ε, σημαντική γιατί λέμε μεταβατική αλλά μεταβατική προς τι ε, σε μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, ναι, αλλά θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετικά ιδιάζουσα συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και επίσης θα είναι μια συνολική συμφωνία η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει την τελική μορφή ε, σχέσης ε, μεταξύ τη Βρετανίας ε, και Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό το άρθρο 50 λοιπόν αναφέρει ρητά ότι πρόκειται για απόσυρση αλλά αυτή η συμφωνία απόσυρσης θα πρέπει να λάβει υπόψη να αναφέρει και τις ε, μελλοντικές ε, ε, σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες μέλη της Ιδίας. Με κάποιο τρόπο λοιπόν αυτές οι μελλοντικέ σχέσεις θα πρέπει να ενσωματωθούν, αλλά εάν ε, προχωρήσει παραπέρα και από την ε, Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου και προχωρήσει παραπέρα ε, που είναι και πολύ πιθανό τότε και, και γίνει ένα είδους συμφωνία ΣΕΤΑ, δηλαδή μεικτή συμφωνίας, τότε αυτό θα σημάνει και επικύρωση από τα κράτη-μέλη μια διαδικασία η οποία ενδεχομένως δεν θα δώσει έτσι κάποια τελικά αποτελέσματα συγκεκριμένα. Ξέρω ότι στις έρευνές σας ε, έχετε συμπεριλάβει και αυτόν τον κίνδυνο. Τον επόμενο μήνα θα υπάρξουν κάποια αιτήματα ε, διευκρίνησης από τη Μεγάλη Βρετανία ε, προς το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με σημεία του άρθρου 50. και καταλαβαίνετε ότι η διαδικασία και αυτή δεν θα είναι πολύ εύκολη. Επίσης, από ό,τι ακούμε εδώ, όταν έρχονται ε, οι εκπρόσωποι της ε, διοίκησης από τη Σκοτία ή από την Ιρλανδία, Καταλαβαίνουμε ότι ε, αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερο προβληματισμό την ε, κατάσταση. Έχουν αρχίσει και συμμετέχουν ε, και σε ακροάσεις, ακροάσεις και του δικαστηρίου και πραγματικά θα πρέπει για την Σκοτία ή για την Βόρεια Ιρλανδία να βρεθεί κάτι ιδιαίτερο το οποίο όμως μπορεί να αποτελέσει ε, συνταγματικό πρόβλημα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένος όσον αφορά ε, το θέμα αυτό ή δεν θεωρείτε ότι είναι ιδιαίτερο πρόβλημα ή ότι θα πρέπει να βρεθούν ιδιαίτερες λύσεις ε, κυρίως όσον αφορά ας πούμε την εσωτερική αγορά. Αν μπορούσατε να μας πείτε λοιπόν κάτι όσον αφορά τη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία ιδιαίτερα. Επίσης το θέμα που αναφέρατε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να ε, υποφέρει από ελλείψεις ε, στην αγορά εργασίας και ο Τζόρτζ προηγουμένως ε, αναφέρθηκε σε αυτό, ότι δηλαδή μπορεί και η αλλαγή της κατάστασης να οδηγήσει και σε αλλαγή διάθεσης, γιατί ενδεχομένως κάποιες διαδικασίες τελικά ε, να μην αποβούν ε, ευεργετικές όσον αφορά το βιωτικό επίπεδο των Βρετανών και ενδεχομένως ε, να υπάρξουν και αντίστροφες μεταναστευτικές κινήσεις λόγω ακριβώς της πτώσης του βιωτικού επίπεδου. Εσείς πιστεύετε ότι όλη αυτή η κατάσταση και όλα τα στοιχεία αυτά ε, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα δεύτερο ε, δημοψήφισμα το οποίο βεβαίως από πολιτικής απόψεως αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζεται. Μήπως θα μπορούσε όμως ε, το τελικό φινάλε να είναι διαφορετικό από αυτό που πιστεύουμε τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά Γκραντ. Πρώτα απ' όλα είπατε ότι η Βρετανική κυβέρνηση ίσως θα μπορούσε να είναι ήπια όσον αφορά τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι παραπάνω όσον αφορά την πρόβλεψή σας αυτή που είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη. Λέει η κυρία Σπινέλη. Ε, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τους ε, ε, Βρετανούς που ζουν εκτός των συνόρων της, Ευρωπαϊκής, της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά και για τους Ευρωπαίους πολίτες που ζουν στην Βρετανία. Δεύτερη ερώτηση, η οποία σχετίζεται με το ίδιο ζήτημα. Τι σημαίνει αυτή η, η ποιότερη προσέγγιση, softer approach, Σημαίνει ότι η, Ευρωπαϊκή, η Βρετανική κυβέρνηση ε, δεν, θα, δεν προτίθεται να είναι καθόλου ήπια με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Πρόεδρος, ε, βλέπω αγαπητοί συνάδελφοι ότι δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο, επομένως να δώσουμε τον λόγο στον Τσάρλς. Να ξεκινήσω με το τελευταίο θέμα που έθιξε η κυρία Σπινέλη. Γνωρίζω πως η κυβέρνηση αυτή την στιγμή εξετάζει το να υπάρχει ένα διαφορετικό σύνολο κανόνων για τους ε, πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα ε, άλλο σύνολο κανόνων ε, για τους πολίτες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν ειδικοί κανόνες για χώρες με του οποίου το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πολύ στενή συνεργασία. Η Αυστραλία, για παράδειγμα, είναι μια τέτοια χώρα. Άρα λοιπόν αυτοί οι κανόνες de facto θα ισχύουν και για τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και για κάποιες άλλες χώρες. Βέβαια είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από τη δεξιά πτέρυγα των συντηρητικών θα διαφωνήσουν. Θα πούνε γιατί ε, είστε κατά των ε, Ινδου, για παράδειγμα, των κατοίκων των ε, πρώην στην Αφρική. Αυτό είναι ρατσισμός. Δεν γνωρίζω βέβαια τι θα συμβεί. Ελπίζω προσωπικά να ε, μην φτάσουν τα πράγματα μέχρι εκεί. Τώρα, ε, πάνω στα σχόλια του Ρίτσαρντ. Ε, νομίζω πως καταρχάς ο Ρίτσαρντ είναι λίγο πιο αισιόδοξο από εμένα για την αλλαγή της κοινή γνώμης. Ελπίζω προσωπικά να έχει δίκιο. Ε, με ρώτησες λοιπόν για την αλλαγή της άποψης των βουλευτών. Αυτή τη στιγμή οι βουλευτές δεν επιθυμούν να μπλοκάρουν το Brexit. Βέβαια αυτό θα αλλάξει να αλλάξει κοινή γνώμη. διότι θα αλλάξει και η, η αντίληψη της ε, κοινωνίας στο ΕΒ Βασίλειο για αυτά τα θέματα. Δεν ξέρουμε βέβαια τι ακριβώς θα συμβεί, εάν θα υπάρξει αυτή η αλλαγή στην ε, κοινή γνώμη, αλλά πιστεύω πως ε, εάν δεν υπάρξει αλλαγή, κάτι που νομίζω είναι κάτι για το οποίο θα ευθύνεται ο τύπος. Ορισμένες εφημερίδες όπως η Daily Mail, η Sun, η Telegraph, η Daily Express είναι φανατικά υπέρ του Brexit, ακολουθούν πολύ σκληρή γραμμή παρά το γεγονός ότι ε, δεν καλύπτουν το 100% του αναγνωστικού κοινού, έχουν όμως πάρα πολύ μεγάλη επιρροή στην κοινή γνώμη. Είναι πολύ δημοφιλείς εφημερίδες. Ακόμα λοιπόν και αν η οικονομία επιδεινωθεί εξαιτία των επιπτώσεων του Brexit, δεν νομίζω ότι αυτές οι εφημερίδες θα βάλουν αυτές τις ειδήσει ε, στην πρώτη σελίδα. Μπορούν να το ε, παρουσιάσουν διαφορετικά, να το πλέξουν, να πούν ότι οι Γάλλοι και οι Γερμανοί μα έκαναν μια πολύ άσχημη πρόταση, η Κομισιόν ε, μα έπαιξε άσχημο παιχνίδι, άλλοι φταίνε για τι για την κακή συμφωνία που έχουμε για, τα, για την επιδείνωση της οικονομία, οικονομίας μας. Βέβαια, πιστεύω σίγουρα πως η βρετανική οικονομία θα υποστεί πλήγμα μετά το Brexit, παρά το ότι έχει κάποια πλέον εκτήματα λόγω της ε, θέσης της. Ε, Μπορεί, για παράδειγμα, να δούμε πως η οικονομία θα αυξάνεται με μεγαλύτερους ρυθμούς από ότι η οικονομία των χωρών που ανήκουν στην Ευρωζώνη, ε, διότι υπάρχουν κάποιες οικονομικές ποινές ε, στις χώρες Ευρωζώνης, τις οποίες, οι οποίες δεν ισχύουν για το Ηνωμένο Αυτό θα επηρεάσει και τις ε, συνομιλίες, τις διαπραγματεύσεις όπως έγινε και την περασμένη εβδομάδα για τη συζήτηση σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και σίγουρα δεν θεωρώ πως, ε, αρκε... πως ε, δεν θα υπάρξουν βουλευτές ε, συντηρητικοί που θα κρατήσουν τα προσχήματα. Μάλιστα πιστεύω πως αρκετοί θα είναι πολύ σκληρής διαπραγματεύσεις και θα ακούσουμε και πολύ σκληρά λόγια για ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω λοιπόν βραχυπρόθεσμα να αλλάξει κοινή γνώμη, μακροπρόθεσμα όμως ποιος ξέρει. Όταν ε, ενδεχομένως δουν οι πολίτες ε, το τίμημα της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό όμως για να γίνει θα περάσει πολύ καιρός. Πιστεύω ότι οποιαδήποτε συζήτηση τέτοιου τύπου για το δημοψήφισμα αυτή τη στιγμή θα δώσει την εντύπωση πως ε, η πλευρά που υποστηρίζει την, ε, το Remain δεν ξέρει να χάνει. Τώρα, διαπραγματεύσεις. Νομίζω πως ε, λίγο καιρό έχουμε. Δεν νομίζω να μας φτάσει από τη στιγμή που στείλει η κυβέρνηση την επιστολή για ενεργοποίηση του άρθρου 50, πρέπει η Κομισιόν να απαντήσει εντό 2-3 μηνών με την μορφή κατευθυντήριων γραμμών. Τότε το Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει την εντολή. Μετά θα περιμένουμε τι γερμανικέ εκλογέ. Θα χρειαστούν ενδεχομένω ένα-δύο μήνε μέχρι να σχηματιστεί κυβέρνηση στη Γερμανία. Θα περάσει λοιπόν ο καιρό και όπω είπατε κι εσεί, η περίοδο για ε, επικύρωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κάποιοι μήνε. Ε, ίσως και λίγο παραπάνω. 14-15 μήνες λοιπόν απομένουν και περνάμε τώρα και σε αυτή τη μεταβατική συμφωνία. Οι Βρετανικές εταιρείε έχουν πει πως χρειάζονται μια τέτοια μεταβατική συμφωνία και πρέπει να το ξέρουν μέχρι ε, την ε, άνοιξη του 2018, έτσι ώστε να πράξουν και αυτοί αναλόγως. Διαφορετικά δεν θα προλάβουν να ε, αλλάξουν τις έδρες των εταιρεών τους κτλ. Αυτό που έχω ακούσει εγώ και αυτό που ξέρω είναι πως δεν μπορείς να κάνεις μια μεταβατική συμφωνία αν δεν ξέρεις τι θε, πού θε να φτάσεις. Πώς μπορείς δηλαδή να υπογράψεις μια συμφωνία χωρίς να ξέρεις τι θέλεις. Και το άρθρο 50 λοιπόν προϋποθέτει διαπραγματεύσεις και αυτή η μεταβατική συμφωνία προϋποθέτει διαπραγματεύσεις, όμως ε, είναι περιορισμένος ο αριθμός εκείνων που θα πρέπει να εξετάσουν όλες αυτές τις λεπτομέρειες και να αποφασίσουν για τις ε, διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό πιστεύω πως θα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί μια μεταβατική συμφωνία. Μετά, κάτι που δεν με ρωτήσατε και είναι πολύ σημαντικό, είναι η νομική βάση. Ίσως βέβαια άλλοι συνάδελφοι γνωρίζουν περισσότερα από μένα, αλλά νομίζω πως υπάρχει διαφωνία σχετικά με τη νομική βάση και τους διακανονισμούς που θα γίνουν. Η νομική βάση του Συμβουλίου, από ό,τι μου είπε ο κ. Ε, είναι ότι όλα μπορούν να γίνουν υπό το άρθρο 50. Οι ψηφοφορίε πλειοψηφία στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, για παράδειγμα, για κύρωση της, ε, του Brexit, ε, είναι έτσι. Όμω, τι γίνεται στην περίπτωση των μελλοντικών διακανονισμών για τι εμπορικέ συναλλαγέ, Αυτές δεν χρειάζονται επικύρωση εθνική. Πρέπει οι εμπειρογνώμονες, οι νομικοί να αποφανθούν για το τι θα γίνει. Επίσης, νομίζω ότι με ρώτησε για τις μελλοντικέ εμπορικές συμφωνίες και τι γίνεται με την ε, ε, επικύρωσή τους. Θεωρώ πως αν η συμφωνία είναι μεικτή, όπως πιστεύω πως θα είναι, μπορούμε να χωρίσουμε τις συμφωνίες σε δύο κομμάτια. Το κύριο τμήμα, το καλό ας πούμε, που είναι αποκλειστικά κοινοτική αρμοδιότητα και θα ε, περάσει πολύ γρήγορα στο στάδιο της επικύρωσης, στο Συμβούλιο, στο Κοινοβούλιο και ε, ένα άλλο τμήμα που είναι εθνική αρμοδιότητα. Εδώ θα μπορούσε να είναι ξεχωριστή συμφωνία η οποία δεν θα είναι καταστροφική, θα είναι ένα μικρό κομμάτι των ε, συμφωνιών. Μετά, με ρωτήσατε εάν θα αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το άρθρο 50, εάν μπορεί να ανακληθεί ή όχι. Αυτό είναι κάτι που συζητιέται και στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή. Και η γενικότερη άποψη εμπειρογνωμόνων, όπω του Λόρδου Κέρ για παράδειγμα, που έχει γράψει βιβλίο για το άρθρο 50, και του κύριου Πύρη, αν δεν κάνω λάθο, αλλά και του κύριου Τούσκ, του πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι ότι εάν αλλάξουν γνώμη οι Βρετανοί μέχρι το καλοκαίρι του 2018, αν πούν για παράδειγμα, όπα για μισό λεπτό, βλακεία κάναμε, τι, τι γίνεται, τότε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει εάν θα ανατρέψει την διαδικασία, εάν θα επιτρέψει δηλαδή στους Βρετανούς να υποχωρήσουν. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όμως σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ε, δώσει κάποια απόφαση για να διευκρινιστεί το ζήτημα. Και η κυβέρνηση ε, του Ηνωμένου Βασιλείου και η πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή θεωρούν πως ε, δεν γίνεται να ανακληθεί ενεργοποίηση του άρθρου 50 γιατί αυτό θα καθυστερήσει για διάφορους λόγους. Δεν πιστεύω λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο. Δύο σημεία τέλος. Ε, Σκοτία. Ναι, υπάρχουν πολλά νομικά ζητήματα με τη Σκωτία, δεν αναφέρθηκα σε όλα από αυτά. Βέβαια, να σας πω πως πράγματι είμαι μέλος της Συμβουλευτική Επιτροπής της Νίκολα Στέρτζον, ε, αμυστή. Δεν επηρεάζει αυτό σε καμία περίπτωση αυτά που σας λέω εδώ. Αλλά να σας πω ότι υπάρχουν ορισμένοι στη Σκωτία που ελπίζουν να μπορεί η Σκωτία να ασκήσει βέτο στην ενεργοποίηση του άρθρου 50. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρουν. Ε, σύμφωνα λοιπόν με ε, αυτούς. Το Κοινοβούλιο της Σκοτίας έχει το δικαίωμα ψηφοφορίας για θέματα ε, που το αφορούν, όπως το Brexit. Υπό κανονικές συνθήκες όμως. Ε, το, τι σημαίνει αυτό, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα έχουν το δικαίωμα να σκίσουν βέτο στο Brexit. Αυτό πιστεύουν αρκετοί νομικοί. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ε, υπάρχουν βέβαια αυτοί που πιστεύουν ότι η Σκοτία θα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τη θέλησή της και σε αυτό ε, στηρίζεται και η κυρία Στέρτζον, ότι θα μπορέσει έτσι να οδηγηθεί σε ανεξαρτησία η χώρα. Εάν τώρα η Σκοτία έχει τη δυνατότητα να αποχωρήσει μεν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά να παραμείνει στην ενιαία αγορά, αυτό είναι διαφορετικό ερώτημα. Υπάρχουν άλλοι κανόνες, ε, είναι πολύ περίπλοκο όμω το ζήτημα για να πατήθει αυτή τη στιγμή. Επίσης, σύνδεση, devolution. Κανείς δεν έχει προτείνει κάτι γι' αυτό μέχρι στιγμής, αλλά ξέρω πως υπάρχουν αρκετές κυβερνήσεις, όπως για παράδειγμα η κυβέρνηση της Ισπανίας, οι οποίες θα επιθυμούσαν να, υπάρχουν, ε, να ισχύουν άλλες προϋποθέσεις για τη σκοτία. Όμω, εάν η Σκωτία, για παράδειγμα, είχε διαφορετικού ε, κανόνε σχετικά με τη μετανάστευση από το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ξέρω δεν βλέπω γιατί να μην γίνεται κάτι τέτοιο, γιατί να μην είναι νομικά εφικτό. Όταν, ας πούμε, ένας Βέλγος πολίτης δουλεύει στη Σκωτία, μπορεί να πάρει έναν ειδικό ε, αριθμό ασφάλισης, ε, σκοτσέζικο, ο οποίος ε, θα, ισχύει μόνο εκεί και δεν θα έχει καμία επίπτωση στο σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Τερέζα Μέη, βέβαια, έχει δηλώσει ότι θα μειώσει δραστικά τον ε, αριθμό της, των μεταναστών που εισέρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο τι μπορεί να γίνει. Υπάρχουν αυτοί που λένε πως οι μετανάστες θα συγκεντρωθούν στη Σκωτία και στο Λονδίνο μόνο και όχι στην υπόλοιπη Μεγάλη Βρετανία και στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Ποια άλλη ερώτηση. Α, ναι. Εάν ε, η κοινή γνώμη θα αλλάξει η άποψη για το μεταναστευτικό όταν θα δει τις επιπτώσεις της επιχειρήσης από τη μείωση της μετανάστευσης. Κοιτάξτε να δείτε, λυπάμαι που το λέω, αλλά η κοινή γνώμη στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι εχθρική προς τη μετανάστευση. Και πολλοί μάλιστα που ψήφισαν να παραμείνει το ΟΒ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά της μετανάστευσης. Έχουν αρνητική γνώμη για τους μετανάστες. Η πλειοψηφία λοιπόν των ε, Βρετανών θεωρεί πως ε, υπάρχουν υπερβολικά πολλοί μετανάστες στη χώρα τους. Τέλος, ε, κύριε Σπινέλη, ρωτήσατε Μάλλον νομίζω πως απάντησα στην ερώτησή σας σχετικά με αυτό που είχατε ερωτήσει. Ναι, ναι, σας απάντησα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, Τζόρτζ. Μπορώ να θέσω επερώτηση για τη μετανάστευση αυτό το τελευταίο που είπες, Charles. Με εκπλήσει το γεγονός ότι κάποιοι υπέρμαχοι του Remain ε, είναι ε, εχθρική ω προς τη μετανάστευση, όπως είπες. Ε, κάνουμε μια διάκριση. Υπάρχουν 2,2-2,3 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες που μένουν ε, στο Ηνωμένο Βασιλείο, περίπου η μισή από την Κεντρική Ευρώπη. Γίνεται μια τέτοια διαφοροποίηση μεταξύ Γερμανών, Γάλλων κτλ. από τη μία και ε, πολιτών τη Κεντρική Ευρώπη από την άλλη. Δεν το ξέρω, να σα πω την αλήθεια. Όμως, από τι δημοσκοπήσει βλέπω ότι πολλοί από του Remainers θα ήθελαν λιγότερη ευρωπαϊκή μετανάστευση Κυρίως αυτό αφορά τους ε, Βουλγάρους και τους Ρουμάνους. Αυτή είναι η δική μου βέβαια ανάλυση. Κάποιο, κάποια τέτοια ε, δυσπιστία αφορά τους ε, κεντρικούς Ευρωπαίους, όμως δεν νομίζω ότι απευθύνεται πολύ, απευθύνεται πολύ προς τους Γερμανούς και τους Γάλλους. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζαμε να μας ε, δώσετε απαντήσεις στα πάντα, αλλά και εσείς ακόμα έχετε ορισμένες ερωτήσεις αναπάντητες. Ελπίζουμε να σημειωθεί πρόοδος από την, την Βρετανική κυβέρνηση για να κατανοήσει περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση σιγά σιγά, γιατί κάποιες φορές ακούμε σχόλια που δείχνουν ότι δεν έχουν καμία ιδέα ε, για το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι είναι εφικτό και τι όχι. Ας ελπίσουμε λοιπόν για το καλύτερο και ότι θα επανέλθετε στο μέλλον για να μας ενημερώσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφοι, θα προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της μέσης διάταξης. Do you want uh, to hear new president? Έχουμε λέ, ε, καινούριο πρόεδρο πλέον, λέει η κυρία Σπινέλη. So, we can... Uh, Ωραία, ας ε, συνεχίσουμε. Έχω ορισμένε ανακοινώσεις σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών. Στην τελευταία συνεδρίαση, στις 21 Νοεμβρίου, οι συντονιστές αποφάσισαν να κάνουν τις εξής συστάσεις ε, προς την Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά το φάκελο για την Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση της ε, Συμμαχίας του Συνασπισμού Ειρήνης και Ελευθερίας, μια νέα επίσημη πρόσκληση θα αποσταλεί σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κόμμα τουλάχιστον ένα μήνα εκ των προτέρων ε, για να υπάρξει ακρόαση των εκπροσώπων της ε, δυνάμει των σχετικών διατάξεων. Σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού 1141 του 2014, οι συντονιστές ε, συνιστούν την κατάρτιση προφορικής ερώτησης με συζήτηση που θα μπορούσε να ακολουθηθεί από μία έκθεση ιδία πρωτοβουλία ε, που θα αποφασιστεί εν ευθέτω χρόνο. Και τέλο, για την αναθεώρηση του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, οι συντονιστέ συνιστούν την κατάρτιση ε, νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας ε, δυνάμει του κανόνου 46 και του άρθρου 225 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εισηγητή ε, που αναφέρεται και έχει εδώ είναι ο Γιώργ Σούπφλιν. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να πάρει το λόγο, βέβαια. Δεν είναι σχεδόν κανείς εδώ. Α, παρακαλώ, θέλετε. Όχι. Εσείς είστε το ο σχεδόν. Εντάξει, θέλουμε ότι εγκρίνονται όλα αυτά. Ας ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Παρά την ε, αυξημένη προβολή και συνάφεια σε σχέση με τομεί που καλύπτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα ε, ουσιαστικά αγνοείται σε μεγάλο βαθμό από τι πλέον πρόσφατε εξελίξει σχετικά με την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων στην νομική, ένωμη τάξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τη μελέτη που έχουμε εδώ μπροστά μα, αυτό ε, ενέχει τον κίνδυνο αντικρουόμενων υποχρεώσεων που θα επιβάλλονται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως μερών ε, της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Χάρτας. Η μελέτη στην οποία αναφέρομαι έχει φέρει τον τίτλο η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας των Δικαιωμάτων και ε, έχει ζητηθεί από το Τμήμα Πολιτικής για τα δικαιώματα των πολιτών και τις ταγματικές υποθέσεις. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο, να καλωσορίσω αρχικά τον ε, ε δόκτωρα Χιούτερ, Σιούτερ, συντάκτη της μελέτης αυτής, που είναι καθηγητή στο Πανεπιστήμιο τη ε, Λουβά και ε, στο πού το Παρίσι. Επίσης είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και μέλος ε, της Επιτροπής Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Αγαπητέ καθηγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαστε να τον πιο σύντομος και περιεκτικός γιατί πολλά μέλη αποχώρησαν και γνωρίζω ότι δεν υπάρχει πολλή χρόνο. Σε πέντε λεπτά θα σας συνοψίσω το περιεχόμενο της μελέτης. Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα ουσιαστικά αποτελεί ένα ε, μέσο το οποίο καταδιώκει τις συνθήκες από την αρχή. Από το 1957, όταν υπήρξε διαπραγμάτευση για την συνθήκη της Ρώμη, από το 1955 μέχρι το 1957, ήδη το Συμβούλιο της Ευρώπης επεξεργαζόταν την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα. Και η επιλογή να μην έχουμε έναν κατάλογο κοινωνικών δικαιωμάτων και να μην υπάρχουν ε, στόχοι κοινωνικής σύγκληση στην αρχική συνθήκη της Ρώμης, ε, ε, προέκυψε ακριβώς από την επίγνωση ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης θα πρέπει να το αναλάβει αυτό και ότι και τα έξι μέλη θα καλύπτονταν και θα δεσμεύονταν από ε, το ίδιο υπόβαθρο κοινωνικών δικαιωμάτων. Όμως αυτό δεν συνέβη στην πράξη. Τα επίπεδα δεσμεύσεων των επιμέλους ε, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικύλουν και το ευρωπαϊκό, το ενωσιακό δίκαιο έχει αναπτυχθεί με τέτοιον τρόπο ε, που έπληξε ε, τα κοινωνικά δικαιώματα με τρόπους που δεν είχαμε προβλέψει από την αρχή. Από τις συνθήκες λοιπόν έχουμε αναφορές που Πρόκειται κυρίω ε, για συμβολικού χαρακτήρα διατάξει, όμω αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα ενίσχυση των δεσμών με αυτό το πολύ ισχυρό μέσο του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Και ξέρουμε όλοι ότι στο Συμβούλιο τη Ευρώπη υπάρχει μια ε, εντυπωσιακή διαδικασία αναζωογόνηση τη Ευρωπαϊκή ε, Κοινωνική Χάρτα, η διαδικασία του Τωρίνο, και ότι υπάρχουν πολύ ψηλέ προσδοκίε για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη διαδικασία με το να, δείχνει μεγαλύτερη, να δείξει μεγαλύτερη βούληση παραπομπής ε, στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα στο έργο της. Αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν ε, αντιμετωπίζει πραγματικά αυτή τη χάρτα ε, στο ίδιο επίπεδο με την Ευρωπαϊκή Συνθήκη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, γιατί αρχικά δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη τα ίδια επίπεδα δέσμευση. Ε, η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι ένα μέσο à la carte. Επιλέγουν δηλαδή τα κράτη-μέλη ποιε διατάξει θα ακολουθήσουν. Υπάρχει λοιπόν μια άνηση σύνδεση με την Χάρτα. Και δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, είναι αρκετά επιφυλακτικό να δώσει την ίδια βαρύτητα στα ε, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα εξαιτία ε, εν μέρη παρανόηση των η ε, του αντικτύπου ε, στα κοινωνικά δικαιώματα στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό όταν υπήρξε η διαπραγμάτευση το 1999-2000 υπήρχε η παραπομπή στην κοινωνική χάρτα αλλά δεν λάμβανε το ίδιο καθεστώς με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάποια δικαιώματα ε, δεν αναφέρονταν, πιο συγκεκριμένα το δικαίωμα στην εργασία και το δικαίωμα στη δίκαιη αμοιβή όπως ξέρουμε, οι κοινωνικές παροχές της Ευρωπαϊκής ε, Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχουν ε, υπονομευθεί όταν ε, τροποποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να ενταχθεί και να συμπεριληφθεί στις συνθήκες του 2007. Και τελικά, και τέλος, δεν υπάρχει ε, ρητή σύνδεση μεταξύ των δύο μερών. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για δύο λόγους. Πρώτον, έχουμε περισσότερα παραδείγματα τώρα των ευρημάτων ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, έναν αναξάρτητο φορέα εμπειρογνωμόνων που παρακολουθεί την εφαρμογή ε, της ε, χάρτας και εντοπίζει σημεία Αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όταν η Σουηδία εφάρμοσε την ε, απόφαση Λαβάλ του 2007, τροποποιώντας ε, την νομοθεσία επισήμανσης, εργασιακά, στα εργασιακά για τις ε, κοινέ συλλογικέ διαπραγματεύσει. Υιοθέτησε λοιπόν απόφαση το 2010 που, όπου, 12 μάλλον, όπου απεφάνθη το δικαστήριο ότι αυτές ε, οι τροποποιήσεις έρχονταν σε αντίθεση με τις απαιτήσεις της ε, κοινωνικής χάρτας. δεν θεωρείται ακόμα ότι ένα κράτος μέλος που συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο ε, επί της αρχής και ύψο φάκτο συνάδει με την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα. Και αυτό αναφέρεται πολύ συγκεκριμένα σε μία ε, υπόθεση ε, της ΣΕΖΕΤΕ εναντί της Γαλλίας σχετικά με τον εργασιακό χρόνο ε, στη Γαλλία, όπου η Επιτροπή ανέφερε ούτε η κατάσταση των κοινωνικών δικαιωμάτων στην ένωμη ε, τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε η διαδικασία κατάρτισης δευτερογενούς νομοθεσίας ε, θεωρείται υπόθεση μόρφωση των ευρωπαϊκών νομικών κειμένων με την χάρτα. Επομένως, διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι προποθέσει αυτέ από τα κράτη-μέλη τη Συμβουλίου τη Ευρώπη, ακόμα και αν αυτό οδηγεί στην Επιτροπή να καταλήξει στο σβέρασμα ότι υπάρχουν ε, αντιθέσει με το νοσιακό ε, δικαίωμα. Και η υπόθεση Λαβάλ και η εφαρμογή στη Σουηδία είναι καλό παράδειγμα. Δεύτερο λόγο που δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση. Στο πλαίσιο τη κοινωνική οικονομική διακυβέρνηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που ουσιαστικά έχει τέσσερι πυλώνε, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, ε, την ενισχυμένη δημοσιονομική εποπτεία που επιβάλλεται ε, στα κράτη-μέλη που επεφολούνται οικονομικής ε, συνδρομής υπό τους ενωσιακούς κανόνες. Ο χρυσός κανόνας ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει, που θα πρέπει να υφετούν τη συνθήκη για την σταθερότητα, συντονισμό και διακυβέρνηση στο πλαίσιο της ΟΝΕ και τέλος Ευρωπαϊκό Μηχανισμό σταθερότητα για την υποστήριξη των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν οικονομικέ δυσκολίε. Σε κανένα από αυτού τους πυλώνε, λοιπόν, δεν συμπεριλαμβάνονται ουσιαστικά τα κοινωνικά δικαιώματα. Παρά τη δέσμευση της Επιτροπής Juncker, πολιτικές καθημερινέ γραμμές που ανακοινώθηκαν τον Ιούλιο του 2014 από τον Πρόεδρο Juncker, να βελτιωθεί η αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου των μέτρων οικονομικής και κοινωνικής διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται αυτό σε έναν βαθμό, αλλά κυρίως εξετάζουμε, μετράμε δηλαδή τον κοινωνικό αντίκτυπο. Δεν συμμορφούμεθα με τα κοινωνικά δικαιώματα. Δεν ελέγχουμε κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση με τα κοινωνικά δικαιώματα. Υπάρχει σημαντική διαφορά. Πρέπει λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, να ενισχύσουμε τον ρόλο της κοινωνικής χάρτας στην ε, ενωσιακή ένωμη τάξη και ε, στην ε, κοινωνικο-οικονομική διακυβέρνηση. Αυτό θα ήταν ένας τρόπος να ενισχύσουμε την νομιμοποίηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μάτια των πολιτών και να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν ε, έχουν αντικρουόμενες υποχρεώσεις από το νοσιακό δίκαιο από τη μία και από την κοινωνική χάρτα από την άλλη και θα επέτρεπε εξέβρεση νέων ισορροπιών ε, μεταξύ της οικονομικής κατάστασης ε, και των υπολείπων ε, πτυχών της ανθρώπινης ζωής. Κλείνουμε με τέσσερις βασικές συστάσεις. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Χάρτα, κοινωνική χάρτα, θα πρέπει να επηρεάσει την ερμηνεία της Χάρτας Μελλοντών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτή τη στιγμή, παρότι έχει ορισμένες τέτοιες διατάξεις, δεν ερμηνεύεται με βάση τις προποθέσει τη κοινωνική Ευρωπαϊκής Επιτροπής Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, κοινωνικών δικαιωμάτων, συγγνώμη. Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα, λοιπόν, δεν τίθεται σε ισότιμη βάση με την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αυτή είναι η πρώτη σύσταση, λοιπόν, κατά βάση. Ελπίζουμε σταδιακά να ληφθεί υπόψη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά την ερμηνεία της ε, Χάρτας των Δικαιωμάτων. Δεύτερον, στις κατευθύνες γραμμές για τις αξιολογήσεις αντικτύπου που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη προβολή της ε, κοινωνικής χάρτας, που αυτή τη στιγμή ε, ελάχιστα παρουσιάζεται, αμεληταία δηλαδή, μέσω της Χάρτας Τεμελών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμω, όπως προείπα, η Χάρτα Θεμελιών Δικαιωμάτων είναι αρκετά επιλεκτική σε ό,τι αφορά τη διαδικασία κοινωνικών δικαιωμάτων και δεν απαραπέμπει στην ομολογία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Μπορούν λοιπόν να βελτιωθούν οι κατευθύνε γραμμέ. Εγώ χαιρετίζω την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2015. Μια διαβούλευση ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2016 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία και χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι εδώ ο κ. Δελαβρίου σήμερα για να μας εξηγήσει περαιτέρω τι έχει κατά νου η Επιτροπή. Ο Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων θεωρώ ότι μπορεί να οδηγήσει στην ενίσχυση των αξιολογήσεων αντικτύπου για να λάβουν υπόψη περισσότερο ε, τα κοινωνικά δικαιώματα βάσει της ε, συνένεση στα τέσσερα στοιχεία του πυλώνα αυτού ίσες ευκαιρίες, καλύτερη συμμετοχή στην αγορά, ε, δίκαιες εργασιακές συνθήκες, ε, επαρκής ε, κοινωνική προστασία και πρόσβαση στις υπηρεσίες. Τρίτη σύσταση. Η Επιτροπή να προάγει την ταυτοποίηση ενός καινού πυρήνα δικαιωμάτων που θα πρέπει να τηρούν και να σέβονται όλα τα κατημέλη. Οι δεσμεύσει ε, των κρατών μελών απέναντι στην κοινωνική χάρτα είναι άνησης. Όμως υπάρχει ανάγκη εναρμόνιση της ε, εικόνας αυτής και να μην έχουμε κράτη-μέλη που έχουν διαφορετικά επίπεδα δέσμευσης που ε, μπορούν να οδηγήσουν σε στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς, ιδίως ό,τι αφορά τον εργάσιμο χρόνο εργασίας. Και καθώς η υλοποίηση είναι προβλέψιμη. Τέλος εδώ και πολλά χρόνια έχουν ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά με την πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή ε, ε, στην, ε, στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και αυτό ήδη περιλαμβανόταν στην λεγόμενη συνθήκη Σπινέλη στη δεκαετία του 1990. και ε, το θέμα των υποαπόσπαση ε, εργαζομένων ε, είχε συζητηθεί και από το Συμβούλιο της Ευρώπης και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και από την ΝΕΟΚΕ. ήταν κάτι επί του οποίου επανειλημμένα το Κοινοβούλιο είχε πει στην, θα έπρεπε να είχε υπογραμμιστεί όπως υπογραμμίστηκε άλλωστε στο ψήφισμα του Φεβρουαρίου 2014. Εγώ ε, μελέτησα τα υπέρ και κατά ε, αυτής της ε, προσχώρησης και το κατά πόσο είναι εφικτό κάτι τέτοιο και συμπεραίνω ότι είναι δύσκολο και ευαίσθητο θέμα και τα συνταγματικά προσκόμματα δεν υπάρχουν όσον αφορά στο εργαλείο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχει ήδη ε, υλοποιηθεί ας πούμε η προσχώρηση ε, στα εργαλεία του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ε, ή της Συνθήκης των Ηνωμένων ΕΕ Εθνών για άτομα με αναπηρίες και επομένως δεν, κατά αυτή την έννοια δεν υπάρχουν προβλήματα διότι η ίδια η Ένωση έχει διατάξεις και λειτουργεί βάσει ιδια η ευρωπαικη ενωση εχει διαταξει παρόμοιων αποφάσεων. Ευχαριστώ πολύ. would like... Πρόεδρος, θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. In Spanish, please. I, I will speak in Spanish. Um, muchas gracias. Σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεσή σας. Πρόκειται για πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εργασία, ενδιαφέρουσα για όλους μας. Ε, έχω ακόμα αμφιβολίες σχετικά με την δυνατότητα που έχουμε να προχωρήσουμε ε, σε αυτό το θέμα. Πολλές φορές άκουσα την κυρία Σπινέλη να αναφέρεται σε αυτόν τον στόχο για λόγους που κατανοώ απαραίτητα σε σχέση και με την ε, ιστορική αναφορά που κάνατε προηγουμένως. Δύο ερωτήσεις έχω να σας υποβάλω. Πρώτον, πιστεύετε ότι η ανάπτυξη του κοινωνικού πυλώνα στην Ευρώπη τώρα ε, βάσει και των σχετικών ε, διακηρύξεων του κυρίου και δηλαδή κάποια μέτρα ε, Βοήθεια ας πούμε του εργασιακού συστήματος στην Ευρώπη, η δυνατότητα ύπαρξης ενός ε, ε, ελάχιστου, ελάχιστου σχετικού εισοδήματος, όχι ιδιού, σε όλες τις χώρες, αλλά ελάχιστο αντιστοίχου ε, σε όλες τις χώρες. Αυτό θα μπορούσε, ας πούμε, ε, να ε, καθοριστεί σε σχέση με την οικονομική κατάσταση κάθε χώρας ή κάποια μέτρα για την ανεργία μακράς διάρκειας η ε, ε, επικοινωνία μεταξύ των κοινωνικών ε, βίων, των βίων ας πούμε των εργασιακών και των κοινωνικών εισφορών των εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη. Όλα αυτά θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ενδυνάμωση της, του κοινωνικού χάρτη, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι τα κεντρικά στοιχεία του χάρτη. Η ερώτησή μου είναι η εξής Πιστεύετε ότι η ανάπτυξη του κοινωνικού πυλώνα γύρω από αυτές τις ιδέες θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανάπτυξη του χάρτη. Δεύτερον, θεωρείτε ότι μπορείτε να προσυπογράψετε τις, ε, στις συστάσεις ε, τις τέσσερις που μας υποβάλατε μία πέμπτη ε, η οποία θα αναφέρεται στο ενδεχόμενο ή επιχειρήσεις σε σχέση με τον κοινωνικό χάρτη και στα πλαίσια των πολιτικών κοινωνικής ευθύνης τους της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης θα μπορούσαν λέω να εντάξουν την ιδέα ότι η κοινωνική, ο κοινωνικός χάρτης και η ολοκλήρωση, η εφαρμογή της από την πλευρά των επιχειρήσεων θα μπορούσε να αναφερθεί σαν ε, ε, μία μέτρηση της, ε, του, της κοινωνικής συμπεριφοράς. Αυτό ε, συμβαίνει και με το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αποτελεί ας πούμε έδαφος επί του οποίου μπορούν να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις ε, κάποια πράγματα και μήπως και ο κοινωνικός χάρτης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μία αναφορά της, ε, της ευθύνης της εταιρικής των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. They Εάν δεν υπάρχουν άλλε ερωτήσεις από τους συναδέλφου, θα ήθελα τότε να κάνω εγώ μερικέ στον ε, καθηγητή Ντεσούτερ στα Ιταλικά. Χωρίς μικρόφωνο η κυρία Σπινέλη. Παρακαλώ. Λοιπόν, ερώτηση. Πώς βλέπω, ε, πώς, γιατί υπάρχει αυτός ο μεγάλος δισταγμός, η επιφυλεκτικότητα ε, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να ενταχθούν ε, στον κοινωνικό χάρτη. Το ρωτάω αυτό και, το, και αναρωτιέμαι μάλιστα γιατί δεν είμαστε σε περίοδο παχιών αγελάδων. Ε, αντιθέτως διανύουμε μεγάλη κρίση κατά την οποία να απομακρύνονται οι, Ευρώπη, οι πολίτες συγγνώμη, από την Ευρώπη και χώρες φιλοευρωπαϊκές ακόμα όπως η Γερμανία και η Ιταλία. Αυτή η απομάκρυνση έχει και κοινωνικό σκέλος ιδιαίτερος ισχυρό και ένα στοιχείο το οποίο ενδεχομένως ε, ονομάζουμε δεξιά ή λαϊκίστικη δεξιά. Εν πάση περιπτώσει ε, υπάρχει αδιαμφισβήτητα ένα κοινωνικό κομμάτι στο οποίο δεν δίνονται απαντήσεις είτε από το κόμμα της Λεπέν είτε ε, από το πολωνικό πυρς, γιατί και εκεί υπάρχει ένα ισχυρό κοινωνικό τμήμα. Μια συνιστόσα κοινωνική πολύ σημαντική. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το θέμα της ε, δημοσιονομικής πειθαρχία που παραμένει ως ε, μοναδικός συνδετικός ιστός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν καταφέρνει να δώσει, να πλουτίσει, να εμπλουτίσει αυτή την πολιτική με μια πραγματική κοινωνική πολιτική. Ε, γιατί δεν πρέπει να ενδιαφερόμαστε μόνο άχα για την δημοσιονομική οικονομική σύγκληση, αλλά να πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και κοινωνικές παραμέτρους. Το αν και Το ρωτώ αυτό, διότι από συνταγματικής απόψεως, δέστε ας πούμε και το παράδειγμα του Ιταλικού Συντάγματος, Εκεί υπάρχει ένα πρώτο τμήμα το οποίο αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου. Και αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα άρχισαν να έρχονται σε μεγάλη σύγκρουση με το νέο άρθρο υπαριθμών 81 το οποίο εντάχθηκε πριν από ε, λίγα χρόνια και που αφορά ε, την δημοσιονομική εξυγίανση. ας πούμε στην Ιταλία το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στην υγεία, η κοινωνική εταιρική ευθύνη στην οποία αναφέρθηκε ο Σάνσος προηγουμένως συγκρούονται εν τέλει με αυτό το άρθρο για την ε, πειθαρχία, τη δημοσιονομική πειθαρχία και επομένως παραμερίζονται δικαιώματα τα οποία είναι θεμελιώδη. Ερωτώ λοιπόν, λέω μάλλον ότι ε, η προσχώρηση στον κοινωνικό χάρτη θα μπορούσε να δώσει μεγάλη ε, όθηση σε κάποιον ο οποίος θα ήθελε να ε, κρατήσει μια ισορροπία ανάμεσα στα δημοσιονομικά και τους προϋπολογισμούς από τη μία και τα κοινωνικά ή θεμελιώδη δικαιώματα από την άλλη. Αυτά θα ήθελα να σας ρωτήσω ε, μάλλον όχι, να ζητήσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι εδώ μαζί μας, εάν θέλει να προσθέσει κάτι. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Okay. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είμαι από την Γενική Διεύθυνση Απασχόληση ε, για επικεφαλή των ε, διεθνών σχέσεων. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με το Συμβούλιο τη Ευρώπη και με την Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Έχουμε συμφέρει επίση ε, στην ενδιαμεσή διαδικασία η οποία προσπαθεί να αναζωογονήσει την κοινωνική χάρτα. Συνεργαζόμαστε επίση και με τον προηγούμενο Επίτροπο Άντορ και με τον τρέχοντα Επίτροπο για να δρομολογήσουμε τις αλλαγές στον κοινωνικό πυλώνα, των πυλώνα των ε, κοινωνικών δικαιωμάτων. Να σας πω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει σε ισχύ μια διαβούλευση η οποία αναμένεται να τελειώσει φέτος. Σε αυτήν την διαβούλευση αναφέρεται ρητά ο κοινωνικός ε, χάρτης και διάφορες άλλες διεθνείς συμβάσεις, όπως παράδειγμα οι συμβάσεις του ΠΟΕ. Η Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει επίσης προσκληθεί για να συνεισφέρει με την παρουσία της στην διαβούλευση. Επίσης το Συμβούλιο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται τη θέση του. Αυτή λοιπόν η διαδικασία διαβούλευσης θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα γίνει μία ε, συνάντηση, ένα συνέδριο απολογισμού 27 Ιανουαρίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ιδιαίτερα η Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων, συνεδρίασαν αρκετές φορές και προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε ε, για ρεαλιστικά θέματα. Πιστεύω λοιπόν πως τα αποτελέσματα της διαβούλευσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, όπως θα δούμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντελαρού. Θα δώσω τώρα το λόγο στον καθηγητή Ντεσούτερ. Θα είμαι σύντομο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω πρώτα στι ερωτήσει σας. Νομίζω πω είναι πολύ βασικά ερωτήματα αυτά που θέσατε. Ακριβώς γιατί σχετίζονται με την εικόνα που έχουν εν μέρει οι πολίτε για ε, την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και το πώς αυτό σχετίζεται με τα κοινωνικά δικαιώματα. Στο στρατόπεδο των ευρωσκεπτικιστών που ολόνα και μεγαλώνει βλέπουμε ένα φόβο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διωγκωθεί και θα εμφανιστεί ένα τεράστιο ευρωπαϊκό κράτος πρόνοιας και υπάρχουν άλλοι που τους λέμε κοινωνικούς σοβινιστές οι οποίοι φοβούνται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαλύσει το κράτος πρόνοιας. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να ε, αναφερθώ στην κοινή γνώμη για την αυτονόητο, αλλά ό,τι και αν κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει σε κάθε περίπτωση να λάβει υπόψη τα κοινωνικά δικαιώματα και να τα θεωρήσει, ε, να τα θεωρήσει ε, πώς όμως περιοριστικά σε αυτό που κάνει καθοδηγητικά, ό,τι κατεύθυνση και ανακολουθήσει ακολουθήσει πρέπει να τα λάβει υπόψη τη και πρέπει να λάβει υπόψη και του περιορισμού που αυτά ε, επιφέρουν στα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, το Σύμφωνο σταθερότητα και Ανάπτυξη είναι καλέ περιπτώσει. Υπάρχει παράγραφος 3,3 τη συνθήκη που αναφέρονται στην δυνατότητα κάποιων παρεκκλήσεων από ορισμένους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους που θα έχουν τα κρατη ε, και αυτό ε, σε εξαιρετικές ε, περιπτώσεις, εξαιρετικές συνθήκες. Ποιες είναι όμως αυτές οι συνθήκες. Όταν παρεκκλίνεις από τους δημοσιονομικούς στόχους, γιατί για να προστατεύσεις τα δικαιώματα των συνταξιούχων, των ανέργων ας πούμε, για να δώσει επαρκή κοινωνική και ασφαλιστική κάλυψη σε αυτές τις ομάδες. Τι ακριβώς θεωρείται εξαιρετικές περιστάσεις. Χρειάζεται λοιπόν ένας μια διευκρίνηση έτσι ώστε η κοινή γνώμη να ε, σταματήσει να ανησυχεί, να καθησυχαστεί και να είναι σίγουρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες των πολιτών. Νομίζω πως ο κύριος Γιούγκερ το έχει κατανοήσει αυτό εις βάθος γι' αυτό και έχει ζητήσει να γίνουν, αυτά, ε, να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι, τα social tests πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση. Πιστεύω λοιπόν πως ε, χρειάζεται μια κοινωνική προσέγγιση η οποία θα είναι βασισμένη στα δικαιώματα τα οποία ε, υπάρχουν, τα οποία είναι κεκτημένα και χωρίς να ξεχνά την ε, κληρονομιά που έχει αφήσει, που έχουν κληροδοτήσει οι προγονείς μας για αυτά τα κοινωνικά δικαιώματα, έτσι ώστε να συνεχίσει το έργο της στο μέλλον. Παίρνω τώρα στην ερώτηση του συναδέλφου, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που με ρωτήσατε, ε, αναφερθήκατε στον πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ως ένα πιθανό διάβλο για να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε την Χάρτα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων περισσότερο στην ευρωπαϊκή πολιτική. Ε, σίγουρα είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουμε. Νομίζω πως είναι βέβαια πολύ νωρίς για να πούμε από τώρα ε, μέχρι πού είναι κανένα να φτάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα ήθελα να κάνω κάποιες προτάσεις. Να πω ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε συμφωνία, συνένεση για τον κοινωνικό πυλώνα εάν βασιστούμε πάνω στο κεκτημένο κοινωνικών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς όπως αναφέρεται στην ε, κοινωνική χάρτα της Ένωσης. Και όπως ορισμένα μέσα του, ε, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ε, για τα κοινωνικά δικαιώματα πρέπει και η κοινωνική χάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι κεντρική στη λήψη αποφάσεων. Πρέπει να δούμε πώς τα κοινωνικά δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών θα ε, έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα ε, στην ε, χάραξη πολιτικής. Και τέλος, έχετε προτείνει κάτι πολύ ενδιαφέρον. στα πλαίσια της προσπάθειας για περισσότερη κοινωνική εταιρική ευθύνη μπορούμε να κάνουμε πολλά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζω πως περιμένει τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν εθνικά σχέδια δράσης που θα βασίζονται πάνω στην έκθεση του 2011 για την κοινωνική εταιρική ευθύνη. Αυτά τα σχέδια δράσης θα πρέπει να λάβουν υπόψη ένα μεγάλο σύνολο δραστηριοτήτων αλλά και τις ε, υποχρε... κοινωνικές υποχρεώσεις των ε, επιχειρήσεων. Πρέπει πιστεύω λοιπόν να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να ε, πιέσουν τι εταιρείε να λαμβάνουν υπόψη του τα κοινωνικά δικαιώματα και τη χάρτα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Γνωρίζω πως υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες προσπάθησαν να συμπεριλάβουν αυτή τη διάσταση. Έχουν γίνει επίσης και άλλες πολλές ε, μελέτες για το πώς η δήλωση των κοινωνικών δικαιωμάτων μπορεί να ενσωματωθεί στις ε, δραστηριότητες της Ένωσης. Όμως ενδεχομένως χρειαζόμαστε ξεχωριστή μελέτη γι' αυτό, γιατί είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση που κάνετε. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τα όσα μας παρουσιάσετε, για την επιχειρηματολογία σας και πιστεύω πως είναι αναγκαίο να συμπεριλαμβάνουμε και αυτή τη διάσταση στην πολιτική και δυστυχώς δεν το σκέφτονται πολύ αυτό, δεν υπολογίζουν πολύ την κοινωνική χάρτα. Να ενημερώσω τώρα για την επόμενη συνεδρίαση η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 8 Δεκεμβρίου από τις 9 μέχρι τις 12.30 το πρωί. Είναι πολύ σημαντικό γιατί θα ψηφίσουμε δύο εκθέσεις. Μετά στις 13 Ιανουαρίου και στις 30 μάλλον Ιανουαρίου και στις 31. 3 με 6,5 και 9 με 12,5. Και εδώ ολοκληρώνεται η συνεδρίαση.